Uh, good morning, dear colleagues. Let's start Καλημέρα ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε σήμερα. Ε, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από ό,τι βλέπω στη μεσηδιάταξη. Ως εκ τούτου μπορούμε να κρίνουμε ότι εγκρίνεται. Καταρχήν, κάποιες ανακοινώσεις. Η Επιτροπή μας και η Επιτροπή ΚΟΝΤ ε, θα ε, ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα καπνικά προϊόντα που θα λάβει η χώρα αυτή η ανταλλαγή απόψεων στις, την Τετάρτη, 12 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί. Στην, ε, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της ε, ΚΟΝΤ έγινε συζήτηση για την εφαρμογή ενός συστήματος για τα χαρακτηριστικά που αφορούν στην καπνική οδηγία και νομίζω ότι με μεγάλη μας χαρά ε, να σας δεχτούμε όλους σας. Δεύτερον, έχουμε ανταλλαγή απόψεων βέβαια σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων ε, για το ε, κέντρο συντονισμού και επίσης και μία συνάντηση μαζί με την ΚΟΝΤ που αφορά στην ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τον ε, ε, μηχανισμό ε, αστικής προστασίας. Πρόκειται για το συντονισμό της αντίδρασης στις καταστροφές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο μηχανισμός ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Όσοι λοιπόν συμμετείχαν κυρίως στην ERCC τον Μάιο καλούνται να συμμετάσχουν και πάλι και πάλι στις 12 Ιουλίου, την Τετάρτη, στις 9 ώρα το πρωί ε, και ε, αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα γίνει από κοινού με την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και θα αφορά στην ε, λειτουργία αυτού του κέντρου συντονισμού. Τα αποτελέσματα ε, θα ληφθούν υπόψη, όπως και ανάλυση των δεδομένων, και θα ληφθούν υπόψη ε, σε σχέση και με την διάμεση αναθεωρήση αυτού του κέντρου που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Την ίδια λοιπόν ημέρα, στις 12 Ιουλίου, στις 12 ε, η ώρα το μεσημέρι, θα γίνει περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της συνάντησης της ΚΟΝΤ, από κοινού με την ΕΝΔΙ και την ΤΕΒΕ, σχετικά με την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, που όπως ανέβρε προηγουμένως, είναι ο μηχανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για για την αστική προστασία. Θα έχουμε και μια έκτακτη συνεδρίαση της ΕΝΒΙ και της ΣΥΤΡΕ, η οποία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 η ώρα μέχρι τις 8.30 το βράδυ στο Στρασβούργο. Και εκεί θα συζητηθούν οι τροπολογίε που κατατέθηκαν για την διαχείριση του ε, χαρτοφυλακίου που αφορά στην Ενεργειακή Ένωση. Σήμερα έχουμε ε, διερμηνία σε 20 γλώσσες ε, και επίσης ε, και έχουμε και ηλεκτρονική ε, μετάδοση της συνεδρίασης. Αν δεν έχετε αντίδραση, τα πρακτικά της 3ης ε, και 4ης Μαΐου, στο τέλος της συνεδρίασής μας, εφόσον δεν θα υπάρχουν αντιρρήσεις, θα υιοθετηθούν, θα κληθούν εγκεκριμένα. Πάμε τώρα στη σημερινή μας συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα είναι οι κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά. Πρόκειται για αναπομπή ε, ο εισηγητής είναι ο κύριος Πότς. Έχετε λοιπόν το λόγο κύριε Πότσο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Ε, κατά τα τελευταία 20 χρόνια ο Ενεργειακός, Ένωση, ο ενεργειακός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφορούσε τα πακέτα τα οποία είχαν σχέση με την μετάδοση, την ε, διανομή, μια νομοθεσία που είχε, είχε σχέση με την ε, μείωση της, ε, των εκπομπών διοξιδίων του άνθρακα, την ανανεώσιμε πηγές ενέργειας και βεβαίω και την ε, ενεργειακή απόδοση. Τον Οκτώβριο του 2014 το, Ενεργειακό, το Συμβούλιο αποφάσισε να χαράξει μέχρι το 2030 τον δρόμο για την ενέργεια και κατόπιν η Συμφωνία των Πορισίων του 2015 επιβεβαίωσε τη βούληση της Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πρωτοπόρα στον αγώνα κατά της κλιματική αναγή. Η μετάβαση λοιπόν στα με τα αποτελεσματικά συστήματα, απαιτεί όμως μια συνοπτική προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συστήσει την ενεργειακή ένεση. Μία από τις βασικές προκλήσεις στον δρόμο προς την οικονομία χαμηλού άνθρακα είναι να υπάρχει η σωστή εφαρμογή της ε, ενέργειας, της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματο. Υπάρχουν ε, κανόνε για το unbundling και αφορούν τον ανταγωνισμό, τις αγορές τη ε, λιανική και της, του χοντρικού εμπορίου Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι τα ηλεκτρικά και ενεργειακά συστήματα θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτα για να αντιμετωπίσουν την όλο και αυξανόμενη ζήτηση για αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας. Βάσει των δεδομένων της Eurostat η ενεργειακή κατανάλωση διπλασιάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια από 14,4% το 2004 σε 28% το 2015. Οι ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας ε, είναι τώρα ανταγωνιστικές σε επίπεδο κόστους και μερικές φορές ε, και πιο φτηνές από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτή η ενεργειακή παραγωγή απασχολεί πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσελκύει περισσότερες επενδύσεις σε πολλούς τομείς και πολλοί τομείς επίσης έχουν περιορίσει τον ορυκτό άνθρακα. Αυτό αντιστοιχεί σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι εντυπωσιακό το ποσό. Εξάλλου όλα αυτά αποτελούν και ένα τμήμα της ενεργειακής ασφάλειας. Οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αυτές ε, ουσιαστικά συμμετέχουν ε, στη ζήτηση του καταναλωτή. Έχουμε νέους παίκτες ε, όπως την τοπική κοινότητα και παράλληλα βλέπουμε ότι αυξάνεται ε, το κόστος. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για τον εφοδιασμό, διότι δεν υπάρχουν νέες επενδύσεις. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο πολλές φορές αντιμετωπίζεται με εθνικά μέτρα. Οι ολοκληρωμένες αγορές χρειάζονται όμως μια ενιαία ρύθμιση και χρειάζονται και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει πάντα ενεργειακή ασφάλεια και δεν θα στρεβλώνονται οι αγορές. Για να αντιμετωπιστούν, να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόγραμμα το πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο. Δύο λοιπόν νομοθετικές προτάσεις αντιμετωπίζουν την, ε, το χοντρικό εμπόριο και το λιανικό εμπόριο και αφορούν ε, τμήματα της ε, αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι βέβαια και μια επιθυμία να υπάρχουν νέες αγορές. Από τότε που οι συντονιστές της Επιτροπής αποφάσισαν να συστήσουν, να συντάξουν μια οδηγία μια γνωμοδότηση για την οδηγία. Έχω και εγώ ε, καταρτήσει τη δική μου έκθεση. Θέλουμε να υπάρξουν τροπολογίες και στον κανονισμό, αλλά βέβαια όλα αυτά θα τα γνωρίζουμε καλύτερα μετά τη σημερινή συνεδρία των συντονιστών. Και ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα να καταθέσουμε τροπολογίες σε αυτό το τμήμα της ε, νομοθετικής διαδικασίας. Αν το κατορθώσουμε αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σε γενικές γραμμές εγώ χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής γιατί υπάρχει όλο και μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε, δεν έχουμε βέβαια σαφείς κανόνες για το λιανικό εμπόριο, για τη λειτουργία των νέων φορέων, όπως επίσης και για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η νομοθετική πρόταση πολύ σωστά βάζει τους κατανοητές στο επίκεντρο της μετάβασης και προσπαθεί να δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι ανανεώσιμες να συμμετέχουν στην αγορά και να υπάρχει περισσότερο περισσότερη περιφερειακή συνεργασία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι της ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής θα επιτυγχάνονται πλήρως τόσο με κανονισμό όσο και με οδηγίες και αυτά πρέπει να τροποποιηθούν σε κάποιο βαθμό. Η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια θα πρέπει να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει ένα ε, βάρος, φορητό βάρος στους καταναλωτές, να αποδοθεί μεγαλύτερη σημασία στην ολοκλήρωση της αγοράς, στην ε, λειτουργία της αγοράς. Για να γίνει αυτό χρειάζονται ίση και όρια ανταγωνισμού για όσους συμμετέχουν στην αγορά. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα δημιουργήσει θεμητό ανταγωνισμό για τη συμμετοχή νέων οντοτήτων όπως είναι οι aggregators ή οι ε, τοπικοί φορείς και παράλληλα δεν θα πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση σε άλλους φορείς. Η ενεργειακή ασφάλεια, ασφάλεια εφοδιασμού δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο, πρέπει να διασφαλίζεται πάντα και η περιφερειακή συνεργασία πρέπει να οθείται από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Αλλιώ θα είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Κατέθεσα περίπου 25 τροπολογίε και προσβλέπω στην αγαστή συνεργασία με του σκιώδει ηγητέ. Το θέμα δεν είναι πολιτική φύσεω, είναι τεχνικό και νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε ουσιαστικά για να επιτύχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Και το τελευταίο είναι, ε, θέλω να υπογραμμίσω, ότι η νομοθεσία για την ενεργειακή αγορά είναι καθοριστική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία τη Ενεργειακή Ένωση. Δύο πυλώνε ε, πρέπει να υπάρχουν. Ο ένα βέβαια είναι προτεραιότητα αυτή τη Επιτροπή. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα βεβαίω ε, έχουν το λόγο οι σκιωδησίτε και συνάδελφοι, εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν. Κυρία Πετικάινεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και στον συνάδελφο κύριο Πόκο για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα στην έκθεση αυτή που μας εξήγησε περί τίνος πρόκειται. Κάποια πράγματα τώρα που νομίζω ότι θα έπρεπε να λάβει υπόψη τη η Επιτροπή μας και για τις τροπολογίες όσον αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα, όλοι γνωρίζουμε ότι η αγορά ηλεκτρισμού περνάει από αλλαγές, εξελίσσεται. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τον άνθρακο και έχουμε πει ότι το 2005 θα έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος ανανόσιμων πηγών ενέργειας. Οπότε για την αύξηση αυτή της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεύτερον, για τα δίκτυα όσον αφορά τη ρύθμιση της παροχής ε, ηλεκτρισμού είναι πράγματα πολύ βασικά ώστε να μπορέσουμε πράγματι να αποφεληθούμε από κάποια ευελιξία. Χρειάζεται ευελιξία για να μπορούμε να αποφελθούμε από αυτά τα δύο ουσιαστικά. Και το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι η αποφυγή του άνθρακα θα έπρεπε να εκφραστεί ποσοτικά και να υπάρξει σαφήνεια όσον αφορά την προτεραιότητα που θα δώσουμε στις ανανεώσιμες. Αλλιώς πάντα θα είναι σε δεύτερη μοίρα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί υπάρχουν τα πυρηνικά, έτσι, οι πυρηνικοί σταθμοί. Και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσαρμόσουμε πόσο θα παίρνουμε από τους πυρηνικούς σταθμούς. Αν λοιπόν δεν αποφασίσουμε πολύ συγκεκριμένα για το τι θα κάνουμε με τις ανανεώσιμες και δεν το εκφράσουμε ποσοτικά, πάντα θα έχουμε τον άνθρακα που θα παρεμβαίνει από την πίσω πόρτα. Και για τις τιμές πρέπει επίσης να φροντίσουμε να υπάρξει μείωση στις τιμές των ανανεώσιμων και σιγά σιγά να κλείσουν οι μονάδες ε, συμβατικών να πούμε ότι θα είναι από τα 50% θα πάει στο 40%, 30% κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι θα κλείσουν οι σταθμοί με συμβατικά καύσιμα. Οπότε, οι καταναλωτές είναι από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά είναι παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά που επίσης μπορούν να παράγουν σημαντικές ποσότητες ηλεκτρισμού και μπορούν να αντικαταστήσουν σε ένα βαθμό τα πυρηνικά. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής παράγει ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρέπει να έχει την ε, προτεραιότητα στην πρόσβαση στις ε, αγορές και αυτό με πολύ καλές τιμές. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε από την ηλιακή ενέργεια και τις ανανεώσιμες γενικότερα. Έπειτα για τεφή δίκτυα. Και εδώ θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Και δεν είναι βέβαια της οδηγίας αυτής, αλλά πρέπει να δούμε το θέμα των super grids, των super δικτύων, και της συνδεσιμότητας. Αν δεν έχουμε ευρωπαϊκή υψηλή τάση, πώς θα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούμε 20% να κερδίσουμε σε ενέργεια από ευφύ δίκτυα και μόνο. Και από αυτό λέει, έχουμε να αποφεληθούμε, χρησιμοποιώντας δηλαδή ευέλικτες πηγές. Σούπερ δίκτυα λοιπόν, ευφύ δίκτυα και ευέλικτη πρόσβαση θα πρέπει να είναι πράγματα τα οποία θα συμπεριλάβουμε στην πρότασή μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Ρής. Ευχαριστώ. Οι σκιώδες για αυτό το θέμα από την ομάδα μας δεν είναι εδώ σήμερα. Οπότε θα σας διαβάσω εγώ τις παρατηρήσεις της. Έχει να πει εξή. Πρώτον, Καλώ ορίζει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πιστεύετε αποτελεί πολύ καλή βάση και ευχαριστεί τον εισηγητή τη γνωμοδότηση, τον κύριο Ποκ. Και να ποια είναι τα θέματα που πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθούν. Πρώτον, για την διευκόλυνση της πρόσβασης των καταναλωτών σε όλες τις διευκολύνσεις της αγοράς ηλεκτρισμού. Επίσης, το θέμα των τιμών πρέπει να απορρέει από ε, διαφάνεια σε μια ανάλυση κόστους και ωφέλους για όλους. Γιατί όταν επιβάλλονται τιμές, μπορούν αυτές να αποτελέσουν και φραγμό για τις εξελίξεις. διότι έτσι δεν υπάρχει προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και δεν υπάρχουν αρκετά κίνητρα για την δημιουργία ηλεκτρισμού. Και αυτό ισχύει κυρίως για τα νοικοκυριά, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ωφέλη. Πρέπει να ληφθούν και αυτά υπόψη όταν αποφασίζουμε πώς θα γίνεται η πρόσβαση από τους καταναλωτές στα δίκτυα. Και τέλος, η κυρία Ποντσέτ λέει ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε τον ρόλο της διασυνδεσιμότητας που είναι πολύ σημαντικό στην αγορά ενέργειας και από πλευράς ασφάλειας ε, ε, προμήθειας αλλά και για να πετύχουμε τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς μας στόχους. Να βελτιώσουμε δηλαδή την απόδοση των ηλεκτρικών συστημάτων και να ε, μην υπάρχει αστάθεια στην εσωτερική αγορά και για τις τιμές, τον καθορισμό τους να συμμετέχουν και οι καταναλωτές. Θα υπάρξουν λοιπόν τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και προσβλέπει σε καρποφόρα συνεργασία με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κλούν είναι επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ τον συντάκτη της νομοδότησης για το έργο του που αποτελεί μια βάση προς Όσον αφορά λοιπόν την αγορά ηλεκτρισμού τώρα, θέλω να αναφερθώ στις τροπολογίες που θα ήθελα να υποβάλω που έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότητα, την απόδοση της ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές και τις ε, καινοτομίες που έχουν να κάνουν με αυτές και τις νέες τεχνολογίες είναι βέβαιο ότι πρέπει να υποστηριχθούν με επιστημονικές μελέτες και άλλες χρηματοδοτήσεις να υπάρξουν επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χρηματοδότηση πρέπει να έχει υπόψη τι γίνεται μακροπρόθεσμα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εκπέμπουν λιγότερες ρηπογόνες ουσίες. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι το θέμα της νομοθεσίας για τα πόβλητα και την κυκλική οικονομία, που στηρίζουμε βέβαια. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία και να λάβουμε υπόψη μας και την υπόλοιπη νομοθεσία, τι λέει για τέτοια ζητήματα, έτσι ώστε η παραγωγή ενέργειας να γίνεται με τρόπο που λαμβάνει υπόψη της όλους τους παράγοντες. Για την αποθήκευση τώρα και πώς θα εξελιχθεί για την νεολική και ηλιακή ενέργεια και πυρηνική. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης στην ε, δικιά μας έκθεση. Το θέμα της επάρκειας στην Ευρώπη, η ασφάλεια εφοδιασμού. Φυσικά είμαστε υπέρ της ειρήνης, είμαι πολιτικός, εννοείται ότι και εγώ θέλω την ειρήνη, αλλά μπορείτε θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Και τέλος να δούμε και το θέμα της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη. Είναι κάτι που δεν συζητιέται πολύ στην ε, Φιλανδία, αλλά στην Ανατολική Ευρώπη, στην Νότια Ευρώπη. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που αναφέρονται στην πρόσβαση σε ενεργειακές πηγές. Ορισμένοι δηλαδή εξαιτίας οικονομικής τους κατάστασης δεν μπορούν καν να έχουν πρόσβαση σε ενέργεια. Έπειτα πρέπει να υπογραμμιστεί περισσότερο ο ρόλος των πολιτών και η συνειδητοποίηση του κόσμου. Και αυτό πρέπει να ενισχυθεί στο κείμενό μας για να συμμετέχουν και αυτοί στις διάφορες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν ε, με τον ενεργειακό κλάδο. Έπειτα για τα δίκτυα τα ενεργειακά, πώς αυτά δημιουργούνται και τα έξυπνα δίκτυα. Εδώ επίσης πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη συνεργασία στην Ευρώπη, ευρύτερη συνεργασία. Και να προχωρήσουμε και με την ιδέα του Energy as a Service. Στις μεταφορές, για παράδειγμα, σήμερα μιλάμε πολύ περισσότερο για την ε, κινητικότητα ως προσφερόμενη υπηρεσία. Το ίδιο να πούμε και για την ενέργεια. Δηλαδή πολύ περισσότερο να τονίσουμε αυτή την έννοια της υπηρεσίας που προσφέρει ενέργεια. Προσβλέπω και εγώ σε καλή συνεργασία με τον ε, συντάκτη γνωμοδότης και με τους κοιόδους ηγητές. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους των Πρεσίνων, λέει ο κύριος Σάντλεκ, ευχαριστώ πολύ για το κείμενο του κυρίου Ποκ, που αποτελεί μια καλή βάση για βελτίωση Θέλω να υπογραμμίσω μερικά πράγματα που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά και μπορούν να καταστήσουν, να βελτιώσουν την γνωμοδότηση αυτή. Μην ξεχνάμε ποιε είναι οι αρμοδιότητε μας. Πρέπει να τις προστατεύσουμε. Και συμφωνώ με προλαλήσατε στην κυρία Κάινεν για παράδειγμα, που λέει ότι πρέπει να στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα για την μείωση των εκπομπών διεξιδίου του άνθρακα την, τον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών και να δούμε ποια είναι τα μέσα που διαθέτουμε που μπορούν να βοηθήσουν για να το πετύχουμε. Είναι σημαντικό επίσης να προσθέσουμε στη γνωμοδότηση αυτή είναι οι μηχανισμοί ικανότητας και πώς θα πετύχουμε τον σημερινό στόχο για τις ε, ενεργειακές αγορές που θα συμπεριλάβουν όλο και περισσότερο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό που δεν βλέπω ακόμα στη γνωμοδότηση, που είναι όμως κεντρικό στο έγγραφο για την Ενεργειακή Ένωση, είναι οι πολίτες η δύναμη αυτή που αποτελούν οι καταναλωτές. Πιστεύω ότι πρέπει το κείμενο να ενισχυθεί περισσότερο σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες και πώς αυτές μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των ε, στόχων και για την κατανομή, να συμμετέχουν, πώς τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά αυτή κατανομής, διανομής μάλλον, ενέργειας. Και η δημιουργία ενέργεια σε μικρή κλίμακα πρέπει να τονιστεί στη γνωμοδότησή μας. Και στο τελικό κείμενο. Οι πολίτες στο μέλλον προφανώς και πρέπει να έχουν ρόλο. Άρα πρέπει να υπογραμμίσουμε το ρόλο των ενεργών πολιτών. Οι κατανοητές είναι σε τρεις κατηγορίες. Η μία είναι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ, αλλά μπορούν να συμμετέχουν για την ολοκλήρωση των δικτύων. Ίσως θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε τον ρόλο και τον ορισμό των ρυθμιστών. των φορέων συγκέντρωσης. Επίσης, να υπάρχουν έξυπνοι μετρητές. Και οι καταναλωτές να μπορούν, εφόσον το ζητήσουν, να έχουν περισσότερες πληροφορίες για τους λογαριασμούς τους. Ε, για την ομάδα τώρα των ενεργών πολιτών πρέπει να ενισχύσουμε τον ενεργό τους ρόλο στη διαχείριση και στο καθορισμό των τιμών της αγοράς. Πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι περισσότερο δραστήριοι σε αυτό το τομέα. Το βασικό, πάση περιπτώσει από τα δικιά μου την πλευρά, είναι η καλή συνεργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί η γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστούμε κυρία Ντονάνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ και σας κύριε Πόκο, για τα έργο σας. Η μεταρρύθμιση της οδηγίας αυτής που έχει να κάνει με κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού είναι η ευκαιρία να υπενθυμίσουμε το ποιοι πρέπει να είναι οι επιθυμητοί στόχοι. Στα πλαίσια λοιπόν της κρίσης μέσα στην οποία βρισκόμαστε, είναι ολοφάνερο ότι μια δημόσια ρύθμιση στις τιμές είναι κάτι αναγκαίο. Διαπιστώνουμε ότι η ελευθέρωση του κλάδου δεν μπόρεσε να διασφαλίσει ασφάλεια εφοδιασμού και σταθερότητα στις τιμές. Εξάλλου η οδηγία αυτή δεν πρέπει να πλήττει την τεχνολογική ουδετερότητα όσον αφορά την επιλογή των πηγών ενέργειας και να πηγαίνουμε προς το όλο από τον ηλεκτρισμό. Και τέτοια τροπολογία θέλω να προσθεθεί στο κείμενο. Τώρα ο εισηγητής έχει δίκιο που θέλει να καταργηθεί το σχήμα για τα δεδομένα. Και όσον αφορά τις διαδικασίες, όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα, που λέγαμε ότι θα αντικαταστήσει τη διαδικασία και τη μορφή των εθνικών αρχών δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε δυσανάλογο βάρος για κάποιες χώρες ε, μέλη που ήδη έχουν κέντρα δεδομένων. Επίσης, συμφωνώ για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις παρά η προσωρινή ρύθμιση των τιμών. Φυσικά πρέπει να περιοριστεί η άνοδος ε, των ε, τιμών του ηλεκτρισμού. Όμως συμφωνώ με τον ε, συντάκτη γνωμοδότησης για το ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, την απόδοση ε, όταν μιλάμε για την αποθήκευση του ηλεκτρισμού. Γιατί η έρευνα κινδυνεύει να δείξει ότι μερικές φορές απειλείται και η ίδια η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των υποδομών αν μειωθεί η ποιότητα, αν πέσει η ποιότητα. Και έπειτα χρειάζεται ένας ελάχιστος ανταγωνισμός ώστε να προωθηθεί η καινοτομία, αλλά ο ανταγωνισμός αυτός δεν θα πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός ώστε να πλήττει τα συμφέροντα των χωρών και των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πεντιτσίνη. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, μέχρι τώρα δουλειά του. Θέλω να σας πω ότι η ενεργειακή πολιτική βασίζεται σε ένα μοντέλο το οποίο έχει ως ε, στόχο ε, να ξεπεράσει την συγκεντρωτική μορφή παραγωγής ενέργειας, να χρησιμοποιούνται περισσότερο ανανόσιμες ψυχές ενέργειας και να περιστεί χρήση του άνθρακα. Συμφωνούμε απόλυτα όσον αφορά τους στόχους της πρότασης. Όσον αφορά βέβαια τους στόχους, διαρωτώ με κατά πόσο είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των διασυνοριακών διασυνδέσεων. Ε, αυτών που επιτρέπουν ε, την πώληση ενέργειας ε, σε χώρες όπως είναι η Ιταλία, που παράγεται όμως ενέργεια, πυρηνική ενέργεια, ας πούμε στη Γαλλία. Τα, οι δύο αυτές χώρες έχουν κάνει επιλογές εκ διαμέτρου αντίθετες, τουλάχιστον όσον αφορά τη μορφή παραγωγής. Όσον αφορά τώρα στους πολίτες και των δύο χωρών, οι Γάλλοι πολίτες πληρώνουν πολύ ακριβά την πυρηνική αυτή ενέργεια που μετά πωλείται πολύ πιο φτηνά στην Ιταλία. Και αυτό εξυπηρετεί στο να διατρείται βέβαια ένα ακριβό σύστημα παραγωγής. Από την άλλη, η Ιταλία πουλάει πάλι στους πολίτες με πολύ υψηλή τιμή. Αυτή η λογική της ε, αγοράς δεν επιτρέπει να συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες και παρότι υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι κανόνες όπως στην Ιταλία και αφορούν στην παραγωγή από ανανόσιμες πηγές, οι πολίτες ε, καλούνται να πληρώσουν την ενέργεια, την ηλεκτρική, πολύ πιο ακριβά από όποιον, οποιοδήποτε άλλο στην Ευρώπη που ε, πληρώνουμε για να διατηρούνται οι μονάδες παραγωγής, για την διάλυσή, του, όταν κρίνονται μη ενεργές. Όλα αυτά οδηγούν στο ότι ε, θα πρέπει αυτές οι πληροφορίες να δίδονται στους πολίτες, γιατί οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι πουδενή σαφής και ευκρινή. Ε, εμεί ε, λοιπόν θα καταθέσουμε και εμεί τροπολογίε για να συμβάλλουμε στην γνωμοδότηση. Άρα, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω στον συνάδελφο Πεντιτσίνη ότι δεν γνωρίζει καλά την κατάσταση στη Γαλλία. Οι Γάλλοι μέχρι τώρα ε, είχαν την ευκαιρία να έχουν τιμές ηλεκτρισμού απόλυτα λογικές. Φυσικά μπορεί να αλλάξει αυτό, αλλά προς το παρόν έτσι είναι. Τώρα, έρχομαι στη συζήτηση για την έκθεση. Συγχαίρω τον συντάκτη γνωμοδότησης, γιατί πραγματικά είναι πολύ σοβαρή η δουλειά που έχει κάνει για ένα θέμα που καθ' άλλο παρά απλό είναι. Αναγνωρίζω ότι η αγορά ηλεκτρισμού πρέπει να είναι πιο ελαστική, γιατί πρέπει να συμπεριλάβουμε τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Συνεπώς χρειάζεται μια δυναμική διαχείριση της κατανάλωσης από τους καταναλωτές, άρα χρειάζεται ευελιξία. Επίσης είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας και τα σημάδια που μας έρχονται από την αγορά για το μακροπρόθεσμο στάδιο. Μπορεί να ενισχυθεί λοιπόν η πρόταση της Επιτροπής για να υπάρξουν συμβάσεις μακροχρόνιες. Όντως χρειάζεται προβλεψιμότητα. Και αν δεν υπάρξουν τέτοιες συμβάσεις μεγάλης διάρκειας, τότε οι επιχειρήσεις μας, οι προμηθευτές μας ενέργειες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Επίσης πρέπει να επιτρέψουμε στις χώρες μέλη να διαθέτουν μηχανισμούς ικανότητας, το είπατε κι εσείς κύριε Σιγητά. Οι μηχανισμοί αυτοί αποτελούν ένα μέσο να διασφαλίσουμε την ε, προστασία εφοδιασμού και πρέπει φυσικά να υποβάλλονται σε κάποιες προϋποθέσεις. Η Κομισιόν έχει πει κάποια πράγματα, λόγω νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο. Και έπειτα υπάρχει και το θέμα της δημιουργίας των ε, τοπικών ε, λειτουργικών κέντρων. Νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή. Αλλά προσοχή, τα κέντρα αυτά δεν θα πρέπει να δυσκολέψουν τους διαχειριστές δικτύων μεταφορών να ελέγξουν την ισορροπία των ηλεκτρικών του συστημάτων. Είναι θεμελιώδες αυτό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι τα αναλυτικά καθήκοντα μπορούν να μεταφερθούν στα κέντρα αυτά, ώστε να υπάρξει καλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς, σύμφωνη, αλλά ό,τι έχει να κάνει με το λειτουργικό, δεν πρέπει να μεταφερθεί. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα φτάναμε να διαχωρίσουμε την ε, ε, λειτουργική απόφαση από τη μία και την ευθύνη από την άλλη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κάποιοι κανόνες επικουρικότητας νομίζω ότι επίσης είναι σημαντικοί εδώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπάλτσο είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις σε σχέση με τις εν λόγω τροπολογίες. Ε, και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μία από αυτές η οποία αφορά την αρχή τη επικουρικότητας ε, Τόσο το Αυστριακό όσο και το Ουγγρικό Κοινοβούλιο έχουν αποστείλει μία αιτιολογημένη έκθεση στον ε, πρόεδρο του Κοινοβουλίου και αυτό γιατί ε, υπάρχει η αίσθηση ότι σε ε, μία σειρά από σημεία η πρόταση προβαίνει σε παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία δημιουργίας ικανοτήτων. Οι εθνικές δεσμευτικέ αρχές θα είχαν, έτσι όπως προβλέπει τώρα η πρόταση, την αρμοδιότητα του να εγκρίνουν τροποντινά τους λόγω μηχανισμούς δημιουργίας ικανοτήτων. αλλά με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ε, καταργούνται κάποιες ε, περαιτέρω δυνατότητες ε, που είχαν τα κράτη-μέλη στην, στην δυνητικέ δυνατότητε των κρατών μελών. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται αυτέ οι αρμοδιότητε στο μέλλον, στον τομέα αρμοδιότητα των κρατών μελών. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μείγμα, το energy mix, εμέσω ε, και πάλι εδώ μειώνεται το πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών. Γίνεται δηλαδή λόγος για ένα ανώτατο όριο ε, των 550 ε, γραμμαρίων ανά κιλοβατόρα, πράγμα που σημαίνει ουσιαστικά ότι οι εγκαταστάσεις δεν θα μπορούν να λειτουργούν με τον τρόπο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς θα καλούνται κάθε φορά να τηρούν τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια. Ούτω ή άλλω και η Συμφωνία του Παρισιού κατέδειξε ότι το κάθε κράτος μέλος φέρει την ευθύνη πλήρωση των λόγων στόχων, αλλά από εκεί και μετά. Εάν δεν είναι σε θέση να επιτύχει την εκπλήρωση αυτών των στόχων με χρήση ορεικτών καυσίμων, τότε ε, ε, ε, η συμφωνία δεν προβλέπει κάτι περαιτέρω σε ό,τι αφορά την μεταβολή του ενεργειακού μείγματο. Δεν προβλέπεται αυτή η δυνατότητα, ωστόσο θα έπρεπε να είναι δυνατό. Από εκεί και μετά θα ήθελα να τονίσω ότι έγινε και μια διαβούλευση σε σχέση με αυτό το ζήτημα στο Αυστριακό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τα επωνομαζόμενα επιχειρησιακά κέντρα, τα οποία ουσιαστικά θα λειτουργήσουν ως αρχές και θα έχουν κάποιους συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας. Αυτά λοιπόν τα επιχειρησιακά κέντρα ουσιαστικά και πάλι θα μειώσουν ε, τις σχετικές αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών μελών. Το κράτος μέλος όμως είναι εκείνο, το εκάστοτε κράτος μέλος ε, ε, είναι εκείνο το οποίο φέρει την ευθύνη ε, για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Εάν λοιπόν ε, ε, τα κέντρα να λάβουν αυτέ τι ευθύνε, δεν θα μπορούν και τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Πότσο ε, για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Η ενιαία αγορά της ενέργειας που να λειτουργεί εύρετμα, αυτό είναι το καλύτερο εργαλείο που μπορούμε να έχουμε για να έχουμε προσιτή ενέργεια. Να διαφυλάξουμε, να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό και να υπάρχει ε, παραγωγή, ικανοποιητική παραγωγή ενέργειας. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, όπως είπε και ο Πάβελ, για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στην προηγμένη τεχνολογία και για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά. Πρέπει να εγγυηθούμε ότι η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια ε, δεν θα είναι ε, ιδιαίτερο βάρος ε, για τους καταναλωτές. Ας έχουμε κατά νου κυρίως τις ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν και την ενεργειακή φτώχεια. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες να κάνουν τη δική τους τη συνδυτή επιλογή για το φορέα που επιθυμούν. Οι ανταγωνιστικές τιμές είναι καθοριστική σημασία για την ευημερία των καταναλωτών και ως εκ τούτου ε, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι καταλητικό για την ε, ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να υπάρχουν ίσοι όρια ανταγωνισμού κυρίως όσον αφορά στους ε, φορείς ε, συγκέντρωση ενέργειας και στις ε, περιφερειακές μορφές συνεργασίας. Να υπάρχουν σαφείς κανόνες. Και τελευταία παρατήρηση σχετικά με την απλούστευση για τις ανώσμες πηγές ενέργειας και για τη συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας. Πρέπει να υπάρχει πιο αποτελεσματική διανομή μέσα από ευφύ συστήματα, να λαμβάνεται υπόψη η φάση προσαρμογής, στα ήδη υπάρχοντα συστήματα, προβλήματα και να είναι πολύ πιο εύκολη με τον τρόπο αυτό και η επιλογή των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντάλη. Thank you. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παύλ Πότσο, τον συγητή Ω προ τα όσα έχει κάνει σε σχέση με αυτή την εγγραμμαδότηση, η οποία νομίζω πω έρχεται στην κατάλληλη χρονική ε, συγκυρία και συνδυάζεται ε, και με το πακέτο για την Ενεργειακή Ένωση, καθώ μα βοηθάει να ξεφύγουμε από τον ε, από αυτή την κεντρική, αν θέλετε, φιλοσοφία όπου έχουμε καταστάσει μεγάλης κλίμακας που βασίζονται στα ορυκτά ε, καύσιμα ε, προς, ε, με μια, προς μια νέα αγορά όπου και οι καταναλωτές και οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ήδη αυτόνομα και να προσαρμόζονται στις, στη ζήτηση της αγοράς παρέχοντας ακριβώς την ενέργεια η οποία χρειάζεται από το σύστημα. Αυτέ λοιπόν οι δυνατότητε ευελιξία σήμερα δεν προβλέπονται στα σημερινά σύστηματα. Το σύστημα λοιπόν στο οποίο στοχεύει ο συγκητής μα οδηγεί ακριβώς αυτήν την νέα αγορά ε, και είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τώρα θα ήθελα να τονίσω ένα-δυο σημείο, ειδικότερα από την περιβαλλοντική οπτική γωνία ε, σε σχέση ειδικότερα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτά είναι τα εξής. Ε, προκειμένου να επιτρέψουμε την ενεργό συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά, ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε βραχυπρόθεσμες αγορές ενέργειας, οι οποίες θα είναι και διαμεθοριακού χαρακτήρα ε, και οι οποίες θα λειτουργούν τόσο προς όφελος των ε, παραγωγών ενέργειας όσο και προς όφελος των καταναλωτών. Ας μην δηλαδή εμένουμε μόνο στα ωφέλη που θα αποκομίσουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές ε, θα αποκομίσουν ωφέλη. Εγώ, καθώς προέρχομαι από τη Μάλτα, ένα πολύ μικρό νησί, πρέπει να τονίσω ότι μια τέτοια νέα αγορά θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη για μικρότερα κράτη-μέλη και φυσικά ε, θα ωφελήσει και ε, τα μεγαλυτερα κρατημέλη στο πλαίσιο δηλαδή της διασυνοριακής εμπορίας ενέργειας που θα λαμβάνει η χώρα. Άρα, όπως ε, ανέφερε και ο Πάβελ, χρειαζόμαστε εδώ περισσότερη ολοκλήρωση των αγορών και μεταρρύθμιση των υφιστάμενων αγορών έτσι ώστε να επιτρέψουμε την εκτεταμένη, ε, την εκτενέστερη ε, συμμετοχή των ανεώσιμων πηγών ε, ενέργειας πράγμα το οποίο έχει ήδη αναφερθεί, αλλά θα μπορούσε να τονιστεί ακόμα περισσότερο. Από εκεί και μετά μου αρέσει το γεγονό ότι γίνεται σαφή αναφορά στην ασφάλεια του ενεργειακού αφοδιασμού. η αγορά δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρί την ασφάλεια. Χρειαζόμαστε και τι δύο πτυχέ προκειμένου να διασφαλίσουμε την ύπαρξη μια αγορά η οποία θα επωφελεί του καταναλωτέ σε γενικότερη βάση. Άρα λοιπόν η ανάληψη και των σχετικών ε, ευθυνών ε, προκειμένου να προβούμε σε την ολοκλήρωση τη ενεργειακή αγορά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίζουμε να τονίζουμε από την πλευρά της και τη Επιτροπή μα. Είμαστε Επιτροπή Περιβάλλοντο, αλλά αφού πρόκειται για κάτι το οποίο μπορεί να αποβεί προ όφελο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και προ όφελο των κατώμελών θα πρέπει να το αναφέρουμε. Τώρα, μ' αρέσουν και αναφορέ που γίνονται στι τοπικέ κοινότητε ενέργεια και στο γεγονό ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ε, καταναλωτέ εκείνοι οι οποίοι ε, δεν συμμετέχουν στα ευρύτερα δίκτυα και συμμετέχουν στι τοπικέ κοινότητε ε, δεν βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την ενεργό συμμετοχή των, των καταναλωτών σε αυτέ τι τοπικέ κοινότητε ενέργεια, ώστε να έχουν ακριβώ τη δυνατότητα να οργανώσουν τι εν λόγω τοπικέ κοινότητε. Επίσης, επιχαίρω το γεγονό ότι γίνεται μια σαφή και εμφαντική αναφορά στου ευάλωτου ε, καταναλωτέ. Όλοι πράγματι οι καταναλωτέ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ε, να ε, λαμβάνουν τι αποφάσει τις, αυτόνομα τις αποφάσεις τους. Δηλαδή συχνά βλέπουμε ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ακριβώς το τι συμβαίνει, ε, ποιος για παράδειγμα ποιο είναι το ύψος της δικής τους ε, παραγωγής ενέργειας ε, που απαιτούν, ποιο, ποια είναι η ενέργεια που ενδείκτηνε να χρησιμοποιούν και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε περισσότερη πληροφορία. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται αναφορά στην ηλεκτρική κινητικότητα, στα ηλεκτρικά οχήματα. Είναι κάτι το, ένας σημαντικός τομέας και καλό είναι να πούμε ότι θα πρέπει να ε, προετοιμάσουμε τη μελλοντική αγορά και για ε, τα ηλεκτρικά οχήματα. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Κλούτση, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλημέρα και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, και εμείς ε, επιχαίρουμε καταρχήν την υποστήριξη ε, της ε, έκθεσης αυτής από την πλευρά δηλαδή, του εισηγητή και από την πλευρά των μελών εδώ της Επιτροπής ε, σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εστιάζει ειδικότερα στους πολίτες στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Επίσης και εμείς έχουμε κοινέ ανησυχίες με τον εισηγητή σε ό,τι αφορά την διευκρίνηση κάποιων ενιών προκειμένου να είναι σαφέστερο το νέο πλαίσιο φορέων για παράδειγμα τι ακριβώς σημαίνουν τοπικές κοινότητες ενέργειας, τι ακριβώς σημαίνουν φορείς συγκέντρηση ενέργειας. Και όλα αυτά βέβαια θα αποβούν και προς όφελος των προσιτών τιμών ενέργειας σε τους καταναλωτές. Γι' αυτό λοιπόν ε, χαιρετίζουμε ε, την, ε, την αναφορά που γίνεται, την πρόταση που γίνεται για διευκρίνηση του, της, της ρύθμισης των τιμών σε έκτακτες περιπτώσεις. Επίσης, θα θέλαμε παρόλα αυτά να ε, ευστήσουμε την προσοχή σας σε μια σειρά από προτάσεις οι οποίες ε, ε, γίνονται και οι οποίες τελικά θα μπορούσαν να μην επωφελήσουν, να μην αποβούν προς όφελος των δικαιωμάτων προ το συμφέρον των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τι αναφορέ που γίνονται στου νέου φορεί αυτού, του φορεί συγκέντρωση ενέργεια, του aggregators, αναφέρθηκαν στη σημερινή συζήτηση επανειλημμένα αυτοί οι νέοι φορεί, γιατί θα κληθούν να αναλάβουν ένα σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση στη ζήτηση και την ευελιξία την οποία θα πρέπει να ενσωματώσουμε στην, στο ενεργειακό μας μείγμα. Δηλαδή η ανταπόκριση στη ζήτηση σήμερα δεν αξιοποιείται πλήρως και γι' αυτό έχουμε προβλέψει και στη δική μας πρόταση μια σειρά από διατάξεις. Αντιλαμβανόμαστε από την πρότασή σας ότι ο εισηγητής ε, ε, θα ήθελε να υπάρχουν κάποιες ρυθμισμένες ε, πληρωμές από την πλευρά των φόρων συγκέντρωσης ενέργειας ό,τι αφορά τα εκάστοτε μέρη. Εμείς στην πρόταση της Επιτροπής έχουμε καταστήσει υπεύθυνα μέρη του balance responsible όπως λέγονται αυτούς τους φορείς συγκέντρωσης ενέργειας γιατί θα πρέπει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς που συμμετέχουν δηλαδή ε, σε αυτήν την ε, ε, στην ευθύνη για την ισόρροπη ζήτηση να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να γίνει μια ρύθμιση σε ό,τι ακριβώς την περίπτωση των φορών γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δεν θα ανταποκρινόμαστε στο πραγματικό κόστος της ανταπόκρισης συζήτηση. Για παράδειγμα, εκείνοι που θα υποφελούνται από την ανταπόκριση στη ε, ζήτηση με βάση τη δική μας ε, πρόταση, ε, στο πλαίσιο για παράδειγμα και της αγωνιστικής πολυσυνέργειας, θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη. Άρα, εάν θέσουμε υπερβολικά υψηλά τον πύχη, όπω προβλέπει η δική σα έκθεση, ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε μια τροχοπέδη στην, ε, στο μηχανισμό ανταπόκριση τη ζήτηση. Ε, γι' αυτό, λοιπόν, εμεί έχουμε προτείνει με αυτόν τον τρόπο τι ε, πληρωμέ μεταξύ aggregators, φορέων συγκέντρωση και προμηθευτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ρόλο που θα αναλάβουν οι αρμόδιοι φορείς ε, των δικτύων διανομής ε, σε σχέση με την ε, συντήρηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ενέργειας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κρατικά μονοπόλια και θεωρούμε πως αυτοί οι φορείς θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν ουδέτερο ρόλο. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και οι εγκαταστάσεις σε ό,τι αφορά το τα οχήματα θα πρέπει να αναπτύσσονται στον, στην ιδιωτική ανταγωνιστική δηλαδή αγορά. Οι ιδιωτικέ επιχειρήσει θα μπορούν να απευθύνονται στου DSOs, αυτού δηλαδή του ε, φορεί ε, των ε, δικτύων διανομή, έτσι ώστε να ε, μπορεί να γίνεται πλήρη αξιοποίηση αυτών των των υποδομών. Ωστόσο, οι DSOs δεν θα πρέπει, θα πρέπει να λαμβάνουν στο ελάχιστο την ευθύνη για τη λειτουργία αυτών των συστημάτων. Οπότε, Εμεί προβλέπουμε τον αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο οι DSOs μόνο σε περίπτωση που υπάρχει αστοχία στην αγορά. Υπάρχει δηλαδή πρόβλημα στη λειτουργία τη αγορά. Ε, με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι οι DSO ε, δια, ε, ε, συγκεντρώνονται στις βασικές τους αρμοδιότητες, δηλαδή την συντήρηση και την επέκταση του δικτύου διανομή. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούν τον ρόλο που είχα μέχρι τώρα, δηλαδή ε, φορέα διευκόλυνση αν θέλετε τη λειτουργία τη αγορά με ουδέτερο χαρακτήρα. Ένα τρίτο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω είναι τα, τα τέλη ε, του switching, switching fees. Μετάβασης. Ε, κάποιες, ε, κάποια κράτη-μέλη όπως η Γαλλία αποφάσισαν να προστατεύσουν πλήρως τους καταναλωτές τους ε, απαγορεύοντας πλήρως τέτοιου είδους τέλη μετάβασης. Αντιλαμβανόμαστε τώρα την πρόταση που κάνετε εσείς ε, και η οποία ουσιαστικά θα οδηγούσε τα νοκο κρατη κράτη-μέλη στο να ανακαλέσουν αυτή την απαγόρευση ε, και ε, στο να επιβάλλουν ουσιαστικά και πάλι τέλη μετάβαση. Αυτό θα, ήταν, ε, θα πρέπει θα ήταν αρνητικό για τους εν λόγω καταναλωτές, γιατί με αυτή την απαγόρευση ουσιαστικά η μετάβαση έγινε πολύ ευκολότερη και η συμμετοχή στον νέο μοντέλο αγοράς. Τέλος, ένα ακόμα σχόλιο που θα ήθελα να κάνω αφορά την ενεργειακή ένδυα, ένα ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε επανειλημμένα στη σημερινή συζήτηση. Είναι πράγματι σημαντικό να πούμε ότι στη δική μας πρόταση έχουμε βρει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα ε, στην ε, δίκαια ανάπτυξη ε, την, και την ισορροπημένη ανάπτυξη της αγοράς αφενός αλλά και την, τις δίκαιες τιμές ενέργειας για όλους. Οπότε γι' αυτό έχουμε προβλέψει για παράδειγμα την υποχρέωση ενημέρωση των καταναλωτών ε, σε ό,τι αφορά τι εναλλακτικέ του δυνατότητε. Ε, και το άρθρο, έτσι όπω το έχουμε διατυπώσει στην πρότασή μα, δίνει μεγάλα περιθώρια ε, ελιγμών στα κράτη-μέλη ω προ το πώ θα εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη διάταξη. Δεν προβλέπει δηλαδή το άρθρο συγκεκριμένα πώ το κάθε κράτο μέλο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει αυτές τις, αυτήν την ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές. Μπορούν ε, να το κάνουν δηλαδή μέσω κάποιου κεντρικού προπολογισμού ή με άλλο τρόπο. Δεν τοποθετούμαστε εμεί το άρθρο προ τον τρόπο αυτό. Όμω, εάν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν αυτήν την εναλλακτική του socialize, τότε θα πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η δυνατότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η μοναδική δυνατότητα θα είναι οι ε, ε, ε, καταναλωτές εκείνοι οι οποίοι είναι πλέον ευάλωτοι, δηλαδή πλέον εκτεθειμένοι σε αποσύνδεση, ακριβώς επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά. Ουσιαστικά δηλαδή η πρότασή σα θα διαιώνιζε αυτό το φαύλο κύκλο, που δηλαδή πλέον ευάλωτοι καταναλωτέ και εκείνοι που υποφέρουν πλέον περισσότερο από τη φτώχεια είναι εκείνοι που επιβαρύνονται περισσότερο. Ο εισηγητής, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, θα ανακεφαλαιώσω και θέλω να αναφέρω να τοποθετηθώ σε κάποια θέματα που ετέθησαν. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που ελέγχθησαν για την πρόσβαση σε ανανεώσιμες, ε, για την παραγωγή μικρής ε, κλίμακας. Ε, πρόκειται για την αναλογικότητα και πρόκειται και για κοινή ευθύνη όσον αφορά την διανομή, χρηματοδότηση, συντήρηση Επίσης, αυτό που παίζει ρόλο είναι και η σταθερότητα των τιμών. Χαίρομαι που ελέγχθη αυτό και χαίρομαι που θα μπορούμε να συνεργαστούμε από αυτού. Επίσης, έγινε λόγος για την, για καινοτομία. Με μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε από αυτού του θέματος και για την αποθήκευση και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, η ενεργειακή φτώχεια ε, σαφώς ε, και είναι προτεραιότητα των σοσιαλδημοκρατών. Θα συνεργαστούμε από αυτού και είναι καλό το ότι η ενεργειακή φτώχεια αυτός ο όρος προέκυψε από τη δική μας την πολιτική ομάδα κατά τη σύνταξη της τελευταίας οδηγίας και συνέβαλα και εγώ σε αυτήν. Όσον αφορά τώρα αυτά που είπαν οι πράσινοι για τους ε, στόχους. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα σίγουρος για το κατά πόσον αυτή η οδηγία είναι στη, στο σωστό σημείο. Μπορούμε βέβαια να συζητήσουμε το ε, κατά πόσο έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε για στόχους. Εδώ πρόκειται για αγορές και θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτά που ρυθμίζει ο κανονισμός για τις αγορές. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να διεκδικήσουμε τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την ε, ανθεκτικότητα όλων των αγορών. Αυτός θα πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος. Η κυρία Ντονάνο αναφέρθηκε στην τεχνολογική ουδετερότητα, στην ασφάλεια της καινοτομίας. Βεβαίως και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Η κυρία Γκροστέτ αναφέρθηκε επίσης σε μηχανισμούς δημιουργίας δυναμικού και υποδομών αυτοί οι μηχανισμοί δεν πρέπει όμως να αντιμετωπίζονται ως ένα είδος συγκαλυμμένων επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Ε, αυτούς τους μηχανισμούς θα πρέπει να τους έχουμε ως ένα είδος μέτρου μετάβασης. Δηλαδή, όταν περνάμε από τεχνολογία έντονης κατανάλωσης του άνθρακα σε άλλη πιο περιορισμένης ε, κατανάλωση του άνθρακα. Αλλά επαναλαμβάνω, όχι να θεωρούμε ότι είναι συγκαλυμμένη επιδότηση ορυκτών καυσίμων. Ευχαριστώ τον κύριο Καπούτο μεταξύ άλλων. Ε, ελπίζω ότι θα δουλέψουμε περισσότερο όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών. Αυτό είναι μια προτεραιότητα των σοσιαλδημοκρατών. Ε, οι αγορές ε, ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως ε, όταν πρόκειται για βραχυπρόθεσμη προσφορά. Σημαντικό μέτρο. Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία που υπήρχε και νομίζω ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί. Όσον αφορά τώρα στο να συγκρίνουμε την ε, πραγματικότητα που υπάρχει στα διάφορα κράτη-μέλη, αυτό που αναφέρατε εσείς, αυτό αποτελεί τη βάση για να υπάρχει μια ισορροπημένη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Όχι μόνο σύγκριση των παλαιών κρατών μελών, αλλά και των αποκαλούμενων σε εισαγωγικά νέων κρατών. Να δούμε τις διαφορές ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο, τα ανατολικά και τα δυτικά κράτη. Όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη, γιατί κατά την άποψή μου, όχι μόνο για μας, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να υπάρχει μια ενοποιητική ολοκληρωμένη στάση. Και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το Κοινοβούλιο αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί το δικό σας το καθήκον είναι η ολοκλήρωση. Όχι να υπάρχει ένα είδος φυγόκεντρων δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ είμαι ανοιχτός για τη συζήτηση υποδειγμάτων και για το πώς ορισμένα μέτρα μπορούν να επηρεάσουν την πραγματικότητα που επικρατεί σε ορισμένα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμβολή σας και ελπίζω να συνεργαστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. 29 Ιουνίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στις 11. Θα ψηφίσουμε την εκτελεστή στις 6 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και περνάμε στο επόμενο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη, που είναι η έκθεση της κυρίας Κοντνέτσνα, ε, Συμφωνεί για την τροποποίηση του πρωτοκόλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε στο Κιγκάλι. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Κονέτσκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρωτόκολλο του Μόντρελ αφορά ουσίες που καταστρέφουν την ε, στιβάδα του όζοντος. Εφτά χρόνια γινόντουσαν διαπραγματεύσεις μεταξύ όλων των μερών και ξεκίνησε από χώρες όπως είναι η Ινδία και η Κίνα που αντιστέκονταν ε, μεν στις αλλαγές αλλά τελικά από την 1η Ιουνίου του 2019 με 20 μέρη τα οποία κατέθεσαν ήδη ε, τη σχετική τεκμηρίωση θα αρχίσει να ισχύει. Τώρα μένει βέβαια η κύρωση από πολλές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία για να δείξει ότι στηρίζουμε αυτή τη συμφωνία και να αποτελέσουμε και παράδειγμα για άλλες χώρες, κυρίως τις αναπτυσσόμενες. Όντω, δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχουν και αλλαγέ αυτές που ξέρουμε τελευταία στις Ηνωμένε Πολιτείε και τις αποφάσεις τη κυβέρνησης, πρόκειται λοιπόν για τους υδροφθοράθρακε. και αυτοί θα συμπεριληφθούν στις ουσίες που καταστρέφουν την ε, στιβάδα του όζοντος. Πριν υπήρχαν ε, οι χλωροφθοράθρακες, τώρα είναι οι υδροφθοράθρακε που του αντικατέστησαν, αλλά εξακολουθούν και αυτοί να χρησιμοποιούνται σε ψυγεία, σε ε, διάφορα υλικά, οικοδομικά κτλ. Και τώρα διαπιστώθηκε ότι ακόμα και οι υδροθωράνθρακες χίλιες φορές παραπάνω καταστρέφουν ε, τη στιβάδα του όζοντο σε σχέση με το διοξίδιο του άνθρακα. Και γι' αυτό και οι ουσίες αυτές θα πρέπει να μειωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Υπάρχει ένα πρώτο στάδιο 2019 και 20. Οι αναπτυγμένες χώρες και οι πιο αναπτυσσόμενες θα μειώσουν τις ε, εκπομπές τους. Το δεύτερο στάδιο 2024-2028 που θα παγώσουν θα παγώσει η παραγωγή τέτοιων ουσιών. Με τη συμφωνία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σηματοδοτήσει τη δέσμευσή της να συνεισφέρει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών όπως έγινε και με το Παρίσι. Είναι πάλι μια πολύ σημαντική συμφωνία, δεσμευτική για να βοηθήσουμε σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας κάτω από τους δύο βαθμούς. Πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και χαίρομαι για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να δεχτεί και να επικυρώσει την τροποποίηση του Κιγκάλη παρά τι ανεξελίξει διαπραγματεύσει για την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε σα παρακαλώ στηρίξτε με την ψηφοφορία σα ε, αύριο αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε. Οι σκιώδε εισηγητέ τώρα έχουν το λόγο. Ο κύριο ε, Φέρια πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για ε, τη δουλειά που έχει κάνει σε αυτό το πολύ σημαντικό φάκελο. Ε, θα ήθελα να αναφέρω ότι στην 28η Σύνοδο Συμβαλωμένων ε, Μερών ε, τη Σύμβαση του Μοντρεόλ που έλαβε χώρα στον Κιγκάλι έγινε μια πρόταση σε ό,τι αφορά την σταδιακή ε, μείωση των ορίων και τη χρήση γενικότερα των υδροφόρων ανθράκων και αντίστοιχη τροποποίηση τη συνθήκη του Μοντρεάλ προκειμένου ακριβώ να τα αποτελεσματικότερα στην κλιματική αλλαγή. Ε, χρειάζεται πραγματικά μια σταδιακή μείωση της χρήσης των υδροφθορανθράκων έτσι ώστε να μειωθεί και η συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή αλλά ε, και, ε, τελικά να οδηγηθούμε στην πλήρη κατάργησή τους. θα πρέπει όμως να γίνει σταδιακά ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, το πρωτόκολλο του Κιγκάλι ε, θα τεθεί σε εφαρμογή όταν θα, έχουν, ε, όταν θα έχει κληρωθεί από τουλάχιστον 20 συμβαλόμενα μέρη. Σε ό,τι αφορά τις σχετικές λοιπόν τροποποιήσεις και προκειμένου να δώσουμε το κίνητρο στις αναπτυσσόμενες χώρες ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να γυρώσουμε αυτήν την τροποποίηση του Κιγκάλη στη Σύμφωνο του Μοντρεάλ προκειμένου να καταδείξουμε τον ηγετικό ρόλο που αναλαμβάνουμε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και προσφέροντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική σε ό,τι αφορά ε, το κλίμα. Ε, ε, ειδικότερα το να αναλάβουμε μια ε, τέτοια στάση ε, είναι πιο σημαντική καθώς ε, οι Ηνωμένε Πολιτείες αποφάσισαν πρόσφατα να μην εφαρμόσουν τις δεμέσεις της Συμφωνίας του Παρισίου. Και στην διάσκεψη κορυφής της Δευτέρας Ιουνίου αναφέρθηκε και σε ψηλότερο επίπεδο η πρόθεση του να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρωτόκολλο του Κιγκάλη. Άρα λοιπόν θεωρώ πως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτή η τροποποίηση του Κιγκάλη να υιοθετηθεί προκειμένου προκειμένου να ανταποκριθούμε στο ρόλο μα σε ό,τι αφορά την ε, καταπολέμηση τη κλιματική μεταβολή και προκειμένου να συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, ε, στο πλαίσιο της ψηφοφορία ε, που θα γίνει αύριο, προκειμένου να εγκρίνουμε δηλαδή αυτή την κύρωση, θα ήθελα να ότι ελπίζω να υπάρξει μαζική υποστήριξη από την πλευρά όλων των συναδέλφων εδώ των μελών της Επιτροπής προκειμένου ή εν λόγω κύρωση από την πλευρά της Ένωσης να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ μιλώ εκ μέρους του Τζο Λάινεν που είναι ο σκιώδης μας ε, για την έκθεση αυτή. Εκ μέρους του λοιπόν Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Κονέτσκα για, την, για το κείμενό της, το οποίο μπορούμε να στηρίξουμε πλήρως. Και δεν μπορούμε να υπογραμμίσουμε αρκετά σήμερα ε, πόσο πολύ προτεραιότητά μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή πρέπει να είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για συμφωνία σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να συμπεριλάβει και τους υδροφθοράθρακες στην συμφωνία αυτή του Μόντρελ στο πρωτόκολλο αυτό. Και τώρα λοιπόν έγινε με η κύρωση και φυσικά και τη στηρίζουμε. Η Επιτροπή αυτή και η Ολομέλεια πρέπει λοιπόν να καταλάβουν ότι έχουν την υποχρέωση να συμφωνήσουν και έτσι να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα στους εταίρους μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μπορούμε να κοιτάξουμε τι έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια με το πρωτόκολλο του Μόντρελ αποτελεί επιτυχία όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και η συμφωνία του Οκτωβρίου στο Κιγκάλι αποτελεί έναν άλλο κρογωνίο λίθο στη διαδικασία αυτή και δείχνει πόσο έχει αναλάβει την υποχρέωση ο κόσμος να προστατεύσει το περιβάλλον και το κλίμα. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα λοιπόν η συμφωνία αυτή του Κιγκάλι για την προστασία του περιβάλλοντος γιατί εφόσον απαγορευτούν οι υδροφθοράνθρακες θα περιορίσουμε και την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη και θα την περιορίσουμε κάτω από τους δύο βαθμούς. Πρέπει λοιπόν η συμφωνία αυτή χωρίς συμβασμούς και χωρίς αλλαγές να περάσει και να μειωθεί η παραγωγή και η κατανάλωση των ε, ουσιών αυτών με συνέπεια. Και οι Ηνωμένε Πολιτείες πρέπει να κυρώσουν τη συμφωνία αυτή προκειμένου να μπορέσει να αρχίσει να ισχύει. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη δικιά στην πλευρά, πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για την κατάργηση των ουσιών αυτών όσο γίνεται πιο γρήγορα λοιπόν προκειμένου να αποτελέσει όντως παράδειγμα στη διεθνή σκηνή. Πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τη δέσμευση να βρει εναλλακτικέ λύσεις. Είναι εφικτό, η οικονομικά είναι επίσης ε, εφικτό και έτσι η Ευρώπη θα έχει ηγετική θέση και θα κρατήσει και τον ανταγωνιστικό της ρόλο στην τεχνολογία αυτή θέρμανσης και ψήξης. Τέλος, η διαδικασία αυτή ε, βοηθάει να προχωρήσουμε και σε άλλες δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος. Οπότε οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες υποστηρίζουμε το σχέδιο σύστασης το οποίο προτείνει η συγκήτρια και θα το υπερψηφίσουμε φυσικά. Ευχαριστούμε λοιπόν τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και περνάμε στον επόμενο μιλητή, η κυρία Ρίση, εκ μέρους της Άλντε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη για να μην επαναλάβω αυτά τα οποία ήδη υπόθηκαν. Δεν είναι επίμαχο το θέμα, για μια φορά. Και για τους φιλελεύθερους, να ξέρετε ότι θα υπερψηφίσουμε, χωρίς ε, ε επιφυλάξεις, χωρίς τροπολογίες και η σκιώδη συζητήτρια μου στηρίζει τα θέματα αυτά και την έκκληση αυτή που λέει ότι πρέπει επιγόντως οι χώρες μέλη να κυρώσουν αυτή τη συμφωνία. Πριν από 25 χρόνια ξεκίνησε η συζήτηση αυτή για το στρώμα όζοντος στο πρωτόκολλο αυτό του Μόντρελ. Διάβασα και έχουν γράψει ειδικοί ότι είχε ε, μειωθεί ε, η τρύπα δηλαδή ήταν στο μέγεθος της Ινδίας τότε. Καλά έκανε και μας υπενθύμησε λοιπόν η συγκέντρια που βρισκόμασταν ε, πριν από 25 χρόνια. Ήταν βέβαια διαφορετικός ο κόσμος, αυτή ήταν η κύρια πρόκληση του κόσμου. Δεν μιλούσαμε τότε για την κλιματική αλλαγή. Χάρη όμως στο πρωτόκολλο του Μότρελ, 98% των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος έχουν απαγορευτεί. Τον Οκτώβριο του 2016 προστέθηκε άλλη μια ουσία με αυτή τη συμφωνία του Κιγκάλη για να καταργηθούν και οι υδροφθοράνθρακες που είναι και αυτά αέρια του θερμοκηπίου 14 φορές πιο δυνατά ισχυρά από το διοτήτιο του άνθρακα και υπάρχουν στα κλιματικά και στα ψυγεία. Οπότε πολύ κάναμε και προσθέσαμε και αυτήν την ουσία στο πρωτόκολλο του Μόντρελ και εφόσον τηρηθεί γρήγορα, γι' αυτό κάνουμε και την έκκληση να κυρωθεί πολύ γρήγορα, θα περιορίσει κατά μισό βαθμό την αύξηση της ε, θερμοκρασίας του πλανήτη. Το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η κύρωση. Επήγαινε να την κάνουν οι χώρες μέλη. και τα η συγκήτρια, μπορούμε να αναρωτηθούμε τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Κέρι ήταν υπέρ. Τι γίνεται όμως με την κυβέρνηση Τραμπ που ξέρουμε ότι αποσύρθηκε και αποσύρεται γενικά από οτιδήποτε έχει να κάνει με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, η τροποποίηση αυτή είναι πολύ σημαντική και θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή. Έχει πληροφορίες για αυτό το θέμα, δηλαδή τι κάνουν οι ΗΠΑ από αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σέικχαουτ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και αντικαθιστώ την κυρία Όκεν που είναι σκιώδης. Έτσι καλώς υπάρχει συνένεση. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια την κυρία Κονέτσκα. Θα την υποστηρίξουμε πλήρως. Βέβαια, γιατί πρόκειται για μια επιτυχία. Πώς δηλαδή η ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό ήταν μία από τις λίγες νομοθεσίες που είχαμε στην προηγούμενη θητεία για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Έγιναν διαπραγματεύσεις σε διεθνές επίπεδο και καταλήξαμε σε επιτυχία στο Κικάλι πέρυσι. Αυτό, συνεπώς, είναι κάτι που πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, γιατί πολλές φορές λέμε πρέπει να κάνει το ένα, πρέπει να κάνει το άλλο. Ε, τουλάχιστον αυτό το έκανε και αποτέλεσε παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση για δράση. Αν λοιπόν αυτή η τροποποίηση εφαρμοστεί πλήρως μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερη θέρμανση του πλανήτη κατά μισό βαθμό. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για καρπούς, για φρούτα στα δέντρα, τα οποία όμως βρίσκονται σχετικά χαμηλά, που εντάξει, αυτή η συζήτηση βέβαια θα πρέπει να ξαναγίνει στο Κιγκάλι για τα πόσο θα έπρεπε να μπει και αυτό μέσα ή όχι. Πάντως, μια ερώτηση έχω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί κυρώνουμε την τροποποίηση αυτή, αλλά μετά πρέπει και να τεθεί σε εφαρμογή η τροποποίηση αυτή. Και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει θέμα διοδότησης εισαγωγών και εξαγωγών στην τροπολογία αυτή, την τροποποίηση αυτή του Κιγκάλι. Στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όμως κάτι τέτοιο δεν εφαρμόζεται πλήρως. Μπορεί κανείς να μιλήσει για ποσοστώσεις, ότι είναι μόνο για τις ε, εισαγωγές, ότι δεν υπάρχει ε, αρκετή αναζήτηση προέλευσης. Αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει πάντως με την εφαρμογή μετά την κύρωση που υποστηρίζουμε πλήρως. Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριο Πετιτσίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κονέτσνα για τη δουλειά της ε, με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Πλέον ε, απαγορεύονται ε, οι ντροφθοράντρακες από τα ψυγεία. Βεβαίως, ας μην ξεχνάμε ότι βλάπτουν κυρίως τα, τις χαμηλές στιβάδες του όζοντος και είναι και πολύ πιο ε, επιβλαβής από το διοξίδιο του άνθρακα. Είμαστε τώρα σε μία παγίδα. Όλο αυτό το θέμα γίνεται και μία ε, αλυσίδα, γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου και την ε, υπερθέρμανση του πλανήτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όποιος ασχολείται με αυτά τα θέματα θα πρέπει να ασχολείται με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η ε, το πρωτόκολλο του Κιγκάλι είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να ζητήσουμε ένα νέο μοντέλο λιγότερης χρήσης του άνθρακα, διότι οι υδροφθοράνθρακες θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από φυσικές ύλες που να είναι και επικερδείς σε όλη αυτή τη διαδικασία της ψήξης και βιομηχανικής ψήξης. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία που πρέπει να την αντράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί για μας προσφέρει τη δυνατότητα να είμαστε στην αιχμή του δώρατος όσον αφορά την τεχνολογία των χαμηλών εκπομπών. Η κυρία Ντορνάνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Κονέτσνα για την ε, παρουσίασή της. Οι υδροφθοράνθακες ε, είναι αέρια του θερμοκηπίου και πρέπει να περιοριστούν. Εδώ να πω δύο θέματα που είναι σημαντικά για μένα. Πρώτον, να σας υπενθυμίσω ότι τα αέρια υδροφθορανθράκων ε, κατ' ουσίαν κρίθησαν ως το υποκατάστατο των χλωροφθορανθράκων που είχαν απαγορευτεί. Απαγορεύτηκαν το 1987 γιατί κατέστρεφαν ε, τη στιφάδα του Όζαντος. Αυτά για τους χλωροφθοράνθρακες. Τώρα και οι υδροφθοράνθρακες όμως αποτελούν ε, απειλή για το πλανήτη και το περιβάλλον γιατί και αυτά ε, συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι αν υποκαταστήσουμε τους υδροφθοράντακες με άλλες ουσίες, αυτές δεν θα πρέπει να συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και όπως και σε πολλές ε, διεθνείς ε, συμφωνίες ε, συμβολική είναι η τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Κιγκάλι. Υπογράφηκε το πρωτόκολλο αυτό από 180 κράτη και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή εδώ έχουμε το αποτέλεσμα μιας διεθνούς ε, συνεργασίας ε, κρατών. Ο κύριος Όουεν. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της ε, που έγινε με πολύ καλό και αποτελεσματικό τρόπο και καταλήγει σε σαφέστατα συμπεράσματα. Νομίζω ότι αυτή η εισηγήση θα μας βοηθήσει στο να κλείσουμε το θέμα ε, όσο πιο γρήγορα γίνεται, το Συμβούλιο να ολοκληρώσει τη δουλειά του στις αρχές του φθινοπόρου και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να καταθέσει την ε, κοινοποίησή της ε, λίγο αργότερα. Όπως ε, ξέρετε, τα κράτη-μέλη προχωρούν με διαφορετική ταχύτητα, αλλά ελπίζουμε ότι στο τέλος θα καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέχρι τον Ιανουάριο του 2019. Ε, ε, Έχουν τεθεί κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά στην στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι αυτού του πρωτοκόλου και των τροποποίησεων. Ε, νομίζω ότι ο Τζον Κέρι ήταν πρωτοπόρος σε αυτά τα θέματα τα προχώρησαν, τα στήριξαν πάρα πολύ, αλλά βέβαια τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία ένδειξη για την ε, δουλειά όλων εκείνων που κάνουν την ε, ε, που εξετάζουν τα θέματα στην πραγματική του διάσταση. Μετά από κάποιες εβδομάδες στην Μπαγκόκ εκεί θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα επίσημα. Τουλάχιστον ε, εγώ αυτή την εντύπωση έχω στη συνεργασία μου με τους ανθρώπους από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τώρα πάμε στην εφαρμογή των τροπολογιών. Σε γενικές γραμμές η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να δεχτεί ε, τις τροπολογίες, να καλύψει αυτά που προβλέπουν όσον αφορά τους υδροφθοράνθρακες, ε, όσον αφορά την αδειοδότηση και την ε, υποβολή αναφορών, πρέπει να κάνουμε κάποιες μικρές αλλαγές για να προσαρμοστούμε ε, στις, ε, στους κείμενους κανόνες. Και όσον αφορά κυρίως την αδειοδότηση, όπως τα ξέρετε, το πρωτόκολλο δεν ορίζει ακριβώς ε, ποιο είναι το σύστημα αδειοδότησης. Βεβαίως εμείς ε, θεωρούμε ότι υπάρχει το σύστημα των ποσοστώσεων το οποίο καλύπτει πλήρως ε, τις προδιαγραφές του συστήματος αδειοδότησης, όπως ακριβώς προβλέπεται στο πρωτόκολλο. Σας ευχαριστώ πολύ. αν να σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τον ε, διάλογο που κάναμε σήμερα και είμαι βέβαια ότι αύριο θα φτάσουμε σε μια, θα επιτύχουμε μια ομόφωνη απόβαση, ούτως ώστε να καταδείξουμε το ρόλο που θέλουμε να λάβουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάσταση των είναι σήμερα στις 5 και αύριο θα γίνει η ψηφοφορία και ελπίζουμε ότι τον Ιούλιο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ε, περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημέρα τη ένταξη, δηλαδή η διασυνορική ρήπανση τη ατμόσφαιρα σε μεγάλη απόσταση και μείωση τη οξύνηση, του ευτροφισμού και του τροποσφαιρικού όζοντο. Ε, ναι. Να σας εξηγήσω λίγο το υπόβαθρο αυτή τη απόφαση του Συμβουλίου. Όλοι γνωρίζετε ε, την ε, ε, ε, όπως γνωρίζουμε υπάρχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις της διασυνοριακής ρήπανσης σε μεγάλη απόσταση στην οικονομία και γι' αυτό η ε, Επιτροπή της Συνεργασίας μεταξύ των 100 μελών και των Ηνωμένων Εθνών έχει ξεκινήσει εργασίες, ε, ε, ξεκίνησε μάλλον εργασίες οι οποίες ε, οδήγησαν το 1979 στην υπογραφή ε, της Σύμβασης για την Διασυνορική Ρήπανση της Ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση. Οχτώ πρωτόκολλα έχουν προσθεθεί έκτοτα και το 8ο πρωτόκολλο του Γκέτεμπορκ είναι εκείνο το οποίο ακριβώς στοχεύει στη μείωση της οξύνωσης του ευτοπλισμού και του τροποσφαιρικού όζοντος θέτοντας ανώτατα όρια για μία σειρά από ατμοσφαιρικούς τρύπους. Το 2012 μία σειρά από τεχνικά παρατήματα αναθεωρήθηκαν προκειμένου να τροποποιηθούν και τα σχετικά οι σχετικέ υποχρεώσει ε, που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη, ειδικότερα προκειμένου να ληφθεί υπόψη και ο μαύρο άνθρακα ή εθάνη. Ε, τώρα λοιπόν θα πρέπει να κυρωθεί αυτό το νέο ε, πρωτόκολλο από τα συμβαλόμενα μέρη τη σύμβαση, προκειμένου να καταστεί δεσμευτικό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρωτόκολλο του Γκέτεμπορκ εφαρμόζεται μέσω της σχετικής ε, οδηγίας και οι τελευταίες ε, τροπολογίες ε, του πρωτοκόλλου θα εφαρμοστούν μέσω της αναθεωρημένης οδηγίας η οποία τέθηκε σε ηχή την 31η Δεκεμβρίου του 2016. Ε, θεωρούμε λοιπόν πως οι τροπολογίες αυτές του πρωτοκόλλου του Γκέντεμπουργκ θα συνεισφέρουν ε, στην επίτευξη ενός υψηλότερου επίπεδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και στη μείωση προφανώς ε, της διαμεθοριακής ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτή την αγώση στο Συμβουλίου και προτείνουμε να συμφωνήσει το Κοινοβούλιο. οπότε, επειδή έχουμε και σχέδιο συζητήσει σε σχέση με αυτό το ζήτημα, θα τους δώσω το λόγο και ξεκινάμε τον κύριο Πολούτσι, νομίζω. Ε, <clears throat> λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ γρήγορα πρόκειται για την επικύρωση των ε, τροπολογιών. Ε, εμείς συμφωνούμε με αυτά με αυτή την επικύρωση πρόκειται για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Γκιότεμπουργκ που πλέον τα όρια είναι πολύ πιο αυστηρά και μπορεί κανείς να επέμβει και σε άλλους ρήπους. Πρόκειται για μια παρέμβαση στη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα στηρίξουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση και αναμένω τη μέρα εκείνη όπου οι πολίτες μας ε, δεν θα απομένουν αυτούς τους ατμοσφαιρικούς ε, ρήπους. Πρόεδρος, από την άλλη δεν έχουμε κάποιον. Κυρία Κονέτσικ, να. Μπορείτε απλώς να πείτε ότι υποστηρίζετε, χρειάζεται να σχολιάσετε. Κύριο Σέικχαουτ. Κάτι Ναι, θα μπορούσα να πω, Πρόεδρε, ότι δεν υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση, αλλά θα ήταν και κάτι το διαφορετικό, αλλά και κάτι το ασφαλμένο. Προφανώς υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση, πρόκειται για εφαρμογή δηλαδή του πρωτοκόλλου και ε, πολύ σωστά είπατε, ε, κυρία Πρόεδρε, ότι ούτω ή άλλω μέχρι το, μέσω των εθνικών ανωτάτων ορίων εφαρμόζουμε αυτό τον περιορισμό. Αλλά είχαμε δει ε, στο, ε, στο, σε σχέση με το προηγούμενο ζήτημα ότι αναλάβαμε ηγετικό ρόλο σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολούθησε ο υπόλοιπο κόσμο. Ενώ αντιθέτω, ε, στο πλαίσιο και των συζητήσεων που έγιναν για την οδηγία των εθνικών ενωτάτων ορίων, η στάση που εθετήθηκε ήταν ότι α μην κινηθούμε πέρα από τα όσα βλέπει το πρωτόκολλο. Ουσιαστικά δηλαδή δεν ανταποκριθήκαμε σε αυτόν τον ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση. Δηλαδή ξεκινάμε με την όλη σύμβαση και τελικά ε, δεν δεν κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, οπότε λίγο είναι απογοητευτικό. Πάντως σε ό,τι αφορά ε, αυτό ε, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, σίγουρα υποστηρίζουμε την έκθεσή σα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, κ. Πεδιτσίνη Εγώ θα πω κάτι κάπως διαφορετικό. Προφανώς ε, και εμείς στηρίζουμε αυτή την τροπολογία. διότι είναι σωστό να αντιμετωπίζεται ο μαύρος άνθρακας ε, ως ατμοσφαιρικός ρήπος. Επειδή όμως μιλάμε για διαμεθοριακή ρήπανση σε παγκόσμια κλίμακα, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτά που είπε ο κύριος Τραμπ. Αν πραγματικά οι ΗΠΑ ε, θεωρούν ότι ο άνθρακας θα πρέπει να είναι πιο ε, σημαντική πηγή εφοδιασμού για την ενέργεια, καταλαβαίνετε ότι εδώ θα μιλάμε για ρήπανση όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά ολόκληρου του κόσμου. Ω εκ τούτου η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει θάρρο και να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία για να δυσχεράνει αυτέ τι εμπορικέ συμφωνίε ανάμεσα στι ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς και αναφέρομαι στο TTIP. Ε, αυτό όμως το έχουν κατά νου οι συνάδελφοι. Από τη μια θέλουν προστασία του περιβάλλοντο, από την άλλη όμω είναι υπέρ του TTIP. Υπάρχουν πάρα πολλές πολυεθνικές που κρύβονται πίσω από αυτές τις συμφωνίες. Ε, δεν πρέπει λοιπόν να τα για αυτά που κάνει ο Τραμπ που φεύγει από τη Συμφωνία των Παρισίων ενώ μόνοι μας στηρίζουμε το TTIP. Αν το κάνουμε αυτό είμαστε οξύμοροι και αντιφατικοί. Ο κύριος Χέντερς εκ μέρους της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που κάνατε για αυτό το θέμα. Εμείς ε, με μεγάλη χαρά βλέπουμε να προχωράει αυτή η απόφαση επικύρωσης, γιατί όπως αναφέρθηκε και στη συζήτηση, η πρόταση της Επιτροπής ανάγεται στο Δεκέμβρη του 2013. Τότε δημοσιεύτηκε ως ε, ένα κομμάτι της δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια, μαζί με άλλες δύο νομοθετικές ε, προτάσεις. Την οδηγία για τα εθνικά όρια ε, και για την οδηγία ε, για τις, τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Προς το παρόν, μόνο τρία μέρη έχουν επικυρώσει τον αθωρημένο πρωτόκολλο συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτή η απόφαση που θα επιτρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επικυρώσει το πρωτόκολλο, αυτή η απόφαση να υιοθετηθεί το συντομότερο δυνατόν. Και αυτό θα ανοίξει τον δρόμο ώστε να ακολουθήσουν και τα κράτη-μέλη. Το ίδιο ισχύει και για όμορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στην Ανατολική Ευρώπη ε, και στην Ασία. Θα ακολουθήσουν και οι χώρες αν δουν ότι προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε λοιπόν αυτή η απόφαση να επιτρέψει την ταχύτατη εφαρμογή του αναθεωρημένου πρωτοκόλλου. Όπως και κάποια κράτη-μέλη και εμεί υπογραμμίζουμε ότι η σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη μπορεί να βοηθήσει ε, στο να περιστούν οι εκπομπέ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρόσφατε μελέτε έχουν καταδείξει ότι η αύξηση τη ατμοσφαιρική τρύπανης σε χώρε όπω η Ινδία και η Κίνα, η αύξηση αυτή επηρεάζει ε, και τι συγκεντρώσει που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μεταφέρονται όλα αυτά τα σωματίδια. Ω εκ τούτου είναι σημαντικό να υπάρχει υπάρχει συνεργασία για διεθνείς ε, συμβάσεις όπως είναι αυτή η σύμβαση για την ε, μεταφορά ρήπων σε μεγάλες αποστάσεις. Ε, Χαιρετίζουμε λοιπόν ε, τη σύστασή σας και ελπίζουμε ε, η ψηφοφορία αύριο να αποβεί θετική. Κάτι μόνο να πω για να τοποθετηθώ σε ένα θέμα ε, που ετέθη από τον κύριο Άικχαουτ σχετικά με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν προχωράνε πιο πέρα στο, συμφών, στο πρωτόκολλο του Γκέτεμπουργκ για τα εθνικά όρια. Πράγματι, αυτό ισχύει για τα έτη μέχρι το 2020. Αλλά η νέα οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια προβλέπει και δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ισχύει όμως αυτή από το 2030 και αυτές οι μειώσεις είναι πολύ πιο αυστηρές από αυτές που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του Γκιούτεμπορκ. Ευχαριστούμε που στηρίζετε αυτό το θέμα. Αύριο θα ψηφίσουμε. Αν θέλετε να καταθέσετε απολογίες, νομίζω σήμερα μέχρι τις 5 και αύριο θα ψηφίσουμε και μετά στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Πρόκειται για μια σειρά ενστάσεων, αντιρρήσεων, βάσει του άρθρου 106. Πρόκειται για τις συνθήκες έγκρισης ενεργών ουσιανδραστικών ουσιών. Έχουμε την ε, θεία μεθοξάμι, το ημίντα κλοπρίτ και την κλωθιανιδίνη. Η κυρία Γκέρλινγκ θα μας εξηγήσει όλα αυτά. Ευχαριστούμε την κυρία Γκέρλινγκ και σας δίνω το λόγο, παρακαλώ, για να μας εξηγήσετε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, δεν θα προσπαθήσω καν να προφέρω τις τρεις αυτές ουσίες, θα τις ονομάσω νεονικοτινοειδή, απλώς. Η πρώτη αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεκτείνει τις, τους περιορισμούς που ήδη ισχύουν όσον αφορά τις δραστικές αυτές ουσίες σε όλες τις καλλιέργειες. Πρώτα απ' όλα με εξέπληξε μια τέτοια απόφαση, καταρχήν γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αμφισβήτηση της του ήδη υπάρχοντος περιορισμού δεν έχει ολοκληρωθεί και επειδή, όπως έχουν πει και άλλοι εδώ τον Ιανουάριο και τον JRC, ότι τα τρέχοντα μέτρα δεν είχαν θετικές επιπτώσεις επί των επικονιαστών. Υπήρχαν αντιρρήσεις λοιπόν ήδη από την προηγούμενη φορά όσον αφορά τις ε, εφαρμοστικές αυτές ρυθμίσεις ότι έχει ξεπεράσει τις αρμοδιότητες της εκτελεστικής Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη τότε. Και τώρα επίσης, και γι' αυτό εξού και η ένσταση αυτή, ο κανονισμός προβλέπει να υπάρξει η έγκριση τέτοιων περιορισμών μόνο εφόσον έχει καταλήξει σε συμπεράσματα βάσει νέας ε, επιστημονικής τεκμηρίωσης και δεν υπάρχουν αρκετά κριτήρια. Επίσης, το παράρτημα 2 λέει ότι απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μία αξιολόγηση κινδύνου να αποδείξει ότι οι δραστικές αυτές ουσίες αποτελούν απαράδεκτο κίνδυνο επί των επικονιαστών. Η ΕΣ έχει πει ότι υπάρχει ψηλός κίνδυνος από τις τρεις αυτές ουσίες, αλλά Ακόμα κι αν βάλουμε στη βάτα τις επικρίσεις που έχουν υπάρξει μέχρι τώρα από τις καθοδηγήσεις που έχουν εκδοθεί για τον πληθυσμό των μελισσών, που έτσι κι είναι ένα επίμαχο θέμα, δεν δικαιολογείται γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αποδείξει ότι πρόκειται για έναν απαράδεκτο κίνδυνο. Ανταυτού αυτές οι προτάσεις γίνονται βάσει ελλείψεων στην γνώση μας. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αποδείξει ότι συμμορφώνεται η απόφασή της με την αρχή της επαγγελματικότητα. Η επέκταση της απαγόρευσης, καλύπτοντας όλες τις καλλιέργειες, θα επηρεάσει πάρα πολύ την γεωργία. Το πρωτόκολλο 2 λέει ότι η δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι κατάλληλη και αναγκαία για να επιτευχθούν οι στόχοι. Σε αυτή την περίπτωση μπορώ να σας πω ότι δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν είναι σαφέ ότι δεν κατάλληλη ρυθμίση αυτή, γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις ε, για τις ε, προϋποθέσεις ότι τα νεονικοτινοειδή αποτελούν απαράδεκτο κίνδυνο και έπειτα ούτε το GRC κατάφερε να αποδείξει τον καταστροφικό αντίκτυπο. Και επειδή η πρόταση αυτή επεκτείνεται σε όλες τις καλλιέργειες, ε, δεν αποδεικνύεται τίποτα τέτοιο και ούτε είναι κάτι αναγκαίο γιατί υπάρχουν άλλα μέτρα που θα μπορούσαν ε, να προταθούν, απαγόρευση κάποιων ε, ε, καλλιεργιών συγκεκριμένων που θα είχαν λιγότερο δραματικές επιπτώσεις στην Γεωργία. Χρειάζεται λοιπόν εκ νέου αξιολόγηση από την ΕΦΣΑ να υπάρξει βεβαιότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και μόνο τότε να υιοθετηθούν νέα μέτρα. Η Επιτροπή πάντως επιμένει ότι αυτή η ρύθμιση είναι καλύτερη. Αλλά εγώ θέλω να τους ρωτήσω γιατί εφόσον το θέμα είναι και στο δικαστήριο δεν περίμεναν. Εκτός από τα επιστημονικά όμως ε, στοιχεία υπάρχει και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι δεν έλαβε υπόψη τις έμεσες συνέπειες της πρότασής της Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι πολύ αρνητικές για το περιβάλλον. Και το πρώτο είναι ο περιορισμός των εναλλακτικών παρασιτοκτόνων που χρειάζονται λιγότερο νερό. Να, ένα αρνητικό. Έπειτα, απώλεια καλλιεργών και αλλαγές. Δεν έχει δώσει σημασία ούτε σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν οι αγρότες δεν μπορούν να έχουν καλλιέργειες γιατί έχουν απαγορευτεί τα προϊόντα δραστικές αυτές ουσίες, δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα τα καταναλώνουμε. Θα τα από το εξωτερικό, από άλλες χώρες, όπου θα έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες δραστικές ουσίες. Οπότε δεν αλλάζει τίποτα. Και ίσως το μεγαλύτερο επιχείρημα είναι ότι μας ε, βάζει, την Επιτροπή μας ε, δηλαδή, σε ενόχους σε αυτήν την ε, προσπάθεια. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα νεονικοτινοειδή, που δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ δεν ασχολούμαστε σε κάτι που πέντε χρόνια πριν λέγαμε στην Επιτροπή μας για περισσότερα χρήματα στην έρευνα για να δούμε γιατί πεθαίνουν οι μέλισσες. Για, θέλω να φτιάξουμε εργαστήρια κτλ. Κανείς δεν μιλάει πια για αυτά. Όλοι μιλούν για τα νεονικοτινοειδή, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι έτσι στρέφουμε την προσοχή αλλού, απλώς και μόνο. Νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στα ουσιώδη, να ασχοληθούμε με το γιατί πεθαίνουν οι μέλισσες και να μην μιλάμε για αυτά τα φυτοφάρμακα για τα οποία δεν υπάρχει καμία απόδειξη. Επίσης, Υπάρχει και μια άλλη ανησυχία, ότι εδώ πρόκειται για μια ιδεολογική συζήτηση. Εγώ έχω ακούσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον του συναδέρφους που πιστεύουν ότι πρόκειται για συμφέροντα των λόμπι, των μεγάλων επιχειρήσεων, αυτοί που είναι κατά των ε, μεγάλων αυτών επιχειρήσεων. Εγώ πρέπει να σας πω ότι μίλησα με πάρα πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις που είναι κατά των ε, παρασιτοκτόνων και συζήτησα μαζί τους, ξέρω ότι θέλουν γενικά τα παριστοκτόνα να αφαιρεθούν από τη Γεωργία, χωρίς όμως να μας λένε τότε τι θα τρώμε στο μέλλον. Και χωρίς να δώσουν αρκετή σημασία στο ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε παριστοκτόνα, αλλά υπεύθυνα να βρούμε τρόπους να διασφαλίσουμε ότι τα χρησιμοποιούμε στη σωστή δόση ότι δεν σπαταλώνται και να ξέρουμε ότι χρειάζεται αυτή η επεξεργασία του σπόρου και να βρούμε έναν τρόπο επεξεργασίας τους που να μην χρειάζεται τα παρασιτοκτόνα αυτά. Με τους ψεκασμούς δεν κινδυνεύουν πάντως οι σπόροι που είναι και αυτή μια ανησυχία κάποιων. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί θέλετε να αφαιρεθούν τα παρασιτοκτόνα από τη Γεωργία. Μπορεί να είναι δικιά σας άποψη, δεν είναι δικιά μου. Και δεν είναι ούτε και η άποψη πολλών, αλλά εσείς υποστηρίζετε αυτήν την προσπάθεια κατακαιρματισμού της πραγματικότητας για να απαγορεύσετε πλήρως κάτι το οποίο είναι κίνδυνο. Τουλάχιστον δεν έχει αποδειχτεί το αντίθετο. Υπάρχουν πάντως ε, πολίτες που ασχολούνται με το θέμα και να ξέρετε ότι σήμερα το βράδυ ε, οργανώνω κάτι που έχει τον τίτλο Evidence Matters, δηλαδή να αποφασίζουμε βάσει στοιχείων, να ξέρουμε τα στοιχεία και όχι να αποφασίζουμε με συναισθηματικά κριτήρια. Κύριε Γκέλινγκ, ευχαριστούμε πολύ, λέει ο η Πρόεδρος. Της 11 πρέπει να πάμε στην Ήτρο, όπω ξέρετε, γιατί έχουμε εκεί να εξετάσουμε το θέμα τη ενεργειακή διακυβέρνηση. Οπότε για τη συζήτηση, ένα λεπτό καθένα παρακαλώ. Γιατί έχω εδώ μακρύ κατάλογο. Πώ θα τα καταφέρουμε. Κάποιοι λένε να εφαρμόσουμε το σύστημα DONT. Ή μπορώ να μην κάνω τίποτα τέτοιο, απλώ να σας ζητήσω να είσαστε επί τη ουσία και να περιοριστείτε στο χρόνο σας. Με τους κοιόδες πρέπει να αρχίσουμε από τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Λένς από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Ε, Εκπροσωπώ σήμερα τον συνάδελφο Πέταγιά, θα ήθελα λοιπόν να πω πως ε, υποστηρίζουμε την αντίληψη αυτή της κυρία ε, κυρίας για τέσσερις βασικούς λόγου ε, λόγους ε, που μου διαβίβασε ο συνάδελφος Καταρχήν η νομική βάση που αξιοποιεί νομική βάση, δηλαδή ένα έγγραφο κατευθυντηριών γραμμών σε ό,τι αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων και τις επιπτώσεις μέλισσες αυτό λοιπόν το έγγραφο καθοδήγηση εδώ και τρία χρόνια απορρίπτεται από την πλειοψηφία των κρατών μελών, οπότε δεν μπορεί να αποτελέσει θεμητή νομική βάση. Ε, και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η ΕΦΣΑ, θα τοποθετηθεί από αυτού του ζητήματο ε, και ε, νομίζουμε πω αυτή η γνωμοδότηση τη ΕΦΣΑ θα είναι η θεμητή νομική βάση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τώρα η Επιτροπή ουσιαστικά προδικάζει την τοποθέτηση τη ΕΦΣΑ. Από εκεί και μετά δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί δεν μα λέει ακριβώ ποιε θα εναλλακτικέ σε ό,τι αφορά την απαγόρευση αυτών των ενεργών ουσιών ε, ε, στα σαχαρότευσλα. Δεν έχουν ε, ληφθεί υπόψη λοιπόν αυτέ οι απόψει. Και τέταρτο ο στόχο είναι το γεγονό ότι εναλλακτικά φυτοφάρμακα για μια σειρά από καλλιέργειε δεν υφίστανται κάτι το οποίο δηλαδή ουσιαστικά δεν θα αποτελούσε μια βελτίωση με την απαγόρευση των σχετικών ενεργών Ουσιαστικά δηλαδή ε, αν χρησιμοποιήσουμε αυξημένα τα υπόλοιπα ε, φυτοφάρμακα ουσιαστικά θα μειώσουμε και την αντίσταση ε, των παθολογικών οργανισμών σε αυτά. Οπότε υποστηρίζουμε από την πλευρά του ΕΛΚ μια διαφορετική άποψη από αυτή της Επιτροπής. η ε, κυρία Ούτελαντ. Ε, αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε ότι πρέπει να συντομεύσουμε λίγο. Θα προσπαθήσω να είμαι πραγματικά συντομότερα. Σας παρακαλώ μην με διακόψετε γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το ζήτημα για την πολιτική μας ομάδα. Θεωρούμε λοιπόν πως υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στην ε, Ευρώπη καθώς βλέπουμε να ε, μειώνεται ο αριθμός των ε, μελισσών μας και υπάρχουν και επιστημονικές εκθέσεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η χρήση χημικών ουσιών είναι ένας από τους λόγους για αυτή τη μείωση του αριθμού των μελισσών. Υπάρχει λοιπόν μια εκτεταμένη επιστημονική συνένεση ότι η έκθεση σε οδεοδικοτινοειδή όπως περιλαμβάνονται σε φυτοφάρμακα έχει ανεδικές επιπτώσεις. Οπότε δεν συμφωνώ με την εισηγήτρια. σε ό,τι αφορά ε, τις ουσίες οι οποίες έχουν απαγορευτεί ήδη το 2013. Ε, σε συνέχεια λοιπόν αυτής της απαγόρευσης ε, θεωρήθηκε πως λόγω τρεις ουσίες αποτελούν πραγματικά ουσίες υψηλού κινδύνου στην Ευρώπη. Οπότε αποφασίστηκε να υπάρξει ε, ε, προσωρινή απαγόρευση. Αλλά έκτοτε έχουμε ουσιαστικά μια, ε, έναν αυξημένο αριθμό επιστημονικών μελετών που επιβεβαιώνουν ότι πράγματι αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για μια σειρά από είδη τα νεοκοτινοειδή και για άλλα είδη, δηλαδή πεταλούδες, έντομα του νερού, ακόμα και για πτηνά. Οπότε έχουμε να κάνουμε εδώ με πάρα πολύ επικίνδυνες ουσίες. Ε, τα απορίσματα λοιπόν ουσιαστικά ενισχύουν τα επιχειρήματα προς ε, ε, υπέρ μάλλον της απαγόρευσης, έστω προσωρινής απαγόρευσης της χρήσης των λόγω ουσιών. Ε, ε, με βάση αυτές τις, ε, αυτά τα νέα επιστημονικά δεδομένα, καλό θα ήταν να προβούν επιτέλους την απαγόρευση των νοικοτινοειδών και καλό θα ήταν να σεβαστούμε πλέον το πόσο επικίνδυνο είναι ο χαρακτήρας αυτών των ουσιών που πραγματικά έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να αποτρέψουμε αυτές τις ζημιές οικοσυστήματα μας. Όλες οι μελέτες καταδεικνύουν ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις για τον αριθμό των μελισσών. Οπότε θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις αρχές της πρόληψης και και υποκατάσταση των ουσιών, αρχές τι οποίες υπογραμμίζουμε ξανά και ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζω επίσης ότι οι πολίτες μας αξιώνουν κάτι τέτοιο. 4,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες συνυπέγραψαν μία έκκληση ε, για την απαγόρευση ακριβώ των νέων νοικοτινοειδών. Θεωρώ λοιπόν ε, πως ε, ε, θα έπρεπε να αναφερθεί και αυτό στη σημερινή ε, εκδήλωση ε, της εισηγήτριας σήμερα. Νομίζω λοιπόν πως εμείς ως μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ της αρχής το ότι μόνο ασφαλή και πραγματικά αποδεδειγμένα ασφαλή χημικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Κυρία γνωρίζετε ότι σας Σέβομαι ε, πολύ και ότι έχω συμφωνήσει και με κάποιες πρωτοβουλίε σα, αλλά σήμερα πραγματικά είμαστε εντελώ αντίθετοι. Δηλαδή ουσιαστικά ε, έχετε ε, πιστεί από τα, το λόμπι της χημική βιομηχανία, το, το οποίο βλέπω εδώ να κάθεται στις τελευταίες σειρέ. Έχω διαβάσει τα όσα έγγραφα μας έχετε διαβιβάσει, αλλά α περάσουμε λίγο στην πράξη. Ε, πώς ε, γίνεται η επεξεργασία των σπόρων με ε, αυτά τα νεονικοτινοειδή. Ε, υπάρχει ένα περίβλημα το, στο οποίο μπαίνουν μέσα, το οποίο περιέχει αυτά τα νεοκοτινοειδή και εφαρμόζεται από τα, στην Κράμβη για παράδειγμα αρχές Αυγούστου έως τον, τον, τα τέλη Απριλίου κάθε μέρα. Δηλαδή, αν τον Δεκέμβριο, για παράδειγμα, υπάρχει ένας επιβλαμής οργανισμός ε, ο οποίος ε, θα ε, βλαστήσει από το έδαφος μου, ξαφνικά θα, μέσα σε τρεις ημέρες θα έχει θανατωθεί. Οπότε, εδώ τι γίνεται. Κάνουμε λόγο συνέχεια για βιοπικιλότητα. Δεν ξέρω. Ε, ουσιαστικά κάνουμε λόγο για μια σειρά από είδη, τα οποία όμω ε, τελικά ε, δείχνουν να εξαφανίζονται όλο και περισσότερο. Ε, εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά τι μέλισσε, ίσω υπάρχουν πιο ειδικοί από μένα, αλλά υπάρχουν μια σειρά από μικροοργανισμοί, τεράστια ποικιλία μικροοργανισμών, οι οποίοι απουσιάζουν πλέον από τα αγροκτήματά μα. Οπότε, αν μα λέτε ότι σε ό,τι αφορά τα ζαχαρότεφλα, για παράδειγμα, ναι, εντάξει, παρατηρούμε ε, το να μην υπάρχει άνθηση των ζαχαροτευτών και εγώ τη ζαχαροτευτών εδώ και 40 χρόνια. Αλλά ε, ούτω ή άλλω τα τρία πρώτα χρόνια ε, ε, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και από εκεί και μετά οτιδήποτε ε, καλλιεργηθεί στα ίδια πάσχει και εκείνο. Ε, όσοι κάθονται τώρα εδώ κάποιοι πρόσωποι, για παράδειγμα της Bayer, ε, ε, γνωρίζουν ότι αυτή η καθημερινή εφαρμογή ε, των παρασυντοκτόνων καθημερινά, ε, μέρα προς μέρα, εβδομάδα προς εβδομάδα, είναι λαθασμένη. Δηλαδή, εγώ λέω ως καλλιεργητής ο ίδιος, ναι, είμαι υπέρ των φυτοφαρμάκων. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε ένα ψεκασμό και να, υπάρχει, να μην υπάρχει πρόβλημα. Ε, τώρα ε, πραγματικά μας λέτε κυρία Γκέρλινγκ ότι δεν υπάρχουν, ε, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε χωρίς αυτές τις ουσίες ζαχαρότητα, πλάι, κράμβι. Ελάτε στο δικό μου αγρότημα να δείτε. Ε, Εντελώ υγιή φυτά, χωρίς να χρησιμοποιούνται νεονικοτινοειδή. Υπάρχουν δεκάδες εναλλακτικέ λύσει. και ουσιαστικά το, το, το, το ζήτημα είναι ότι υπάρχει εναλλακτικό προϊόν εδώ. Άρα λοιπόν τι κάνουν. Οι μεγάλε επιχειρήσει ουσιαστικά προσπαθούν να στήσουν πιέσει στην Επιτροπή μα, ώστε να μπορούν σε δύο χρόνια να ε, συνεχίσουν τη χρήση των ελόγων προϊόντων ε, και μέσα σε δύο-τρία χρόνια να έχουν αναπτύξει αναλυτικά προϊόντα τα οποία μπορούν να πουλήσουν. Οπότε ε, μην του κάνετε τη χάρη. Γιατί αν θέλετε να μην υπάρχουν ε, τέτοιου είδους ουσίες ε, στα γλύματα στο μέλλον για τα παιδιά μας, τότε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορεί από το χέρι μας για να απομακρύνουμε αυτό το δηλητήριο από τις καλλιέργειες μας. Ε, τώρα εγώ σας έδωσα τρία λεπτά και παραπάνω. Εντάξει, δεν πειράζει, αλλά δεν είναι καλό παράδειγμα για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Η κυρία Κονέτσνα, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, διότι εκ μέρους ε, της ε, ομάδας ε, Να πω το εξή. Κατανοούμε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να προτείνουν ό,τι θέλουν. Αλλά ξέρετε, εμεί ήμασταν πολύ προσεκτικοί για αυτά που είπαμε σχετικά με τους παραγωγούς των νεοκοτινοειδών και των αγροτών. Αν δεν έχουμε τις μέλισσες, τι, μιλάμε, δεν θα υπάρχει γεωργία. Και τα νεονικοτονοειδή έχει αποδειχθεί ότι ε, καταστρέφουν, εξαφανίζουν τις μέλισσες. Και όταν θα εξαφανίσουμε όλα αυτά τα ίδια από το οικοσύστημα, θα έχουμε ένα απόλυτο τίποτα. Και τότε όλοι μας θα εκπλαγούμε γιατί τίποτα δεν θα μπορεί να μας βοηθήσει. Η Google λοιπόν ποτέ δεν θα στηρίξει τέτοιου είδους ε, αντιρρήσεις ε, που απειλούν το οικοσύστημα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Αν μπορούμε να κάτι να αμυνθούμε, ας το κάνουμε, γιατί αυτή είναι η μόνη ευκαιρία που έχουμε να ε, προστατεύσουμε την επόμενη γενιά, όχι μόνο των μελισσών, αλλά όλων των όντων του πλανήτη. Κυρία Πρόεδρε, εγώ μιλώ εξ ονοματός μου λέει η κυρία Μούλερ και όχι εκ μέρους ε, του σκιώδης ε, εισηγητή ε, της άλδε. Συμφωνώ με την κυρία Γιόλινγκ. Ρωτώ τον κύριο Φλόρεντ, εσείς τι κάνετε με τα αγροκτήματά σας, τα καλλιεργείτε βιολογικά, έχετε εναλλακτικά προϊόντα. Για μένα, ξέρετε, αυτό που έχει σημασία είναι να επαναξιολογήσουμε την απαγόρευση. υπάρχει πλέον αυτή η επαναξιολόγηση, Μάλλον, η απαγόρευση ισχύει εδώ και τρία χρόνια, αλλά δεν υπάρχει ακόμα επαναξιολόγηση και πρέπει να περιμένουμε. Το έγγραφο B-Guidance ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ούτε αυτό το έχουμε ακόμα στα χέρια μας και τα κράτη-μέλη δεν το έχουν αναγνωρίσει έτσι και αλλιώ. Με βάση λοιπόν αυτά που γνωρίζω, δεν υπάρχει εναλλακτικό μέτρο και εναλλακτική ουσία. Και αυτά που χρησιμοποιούνται ως νέα τεχνολογία, ούτε και αυτά έχουν κριθεί αποτελεσματικά. Ε, εγώ λοιπόν θα ήμουν πολύ προσεκτική. Πρέπει να σας πω ότι ε, δεν ε, έχω δει κάποια συγκεκριμένη μελέτη η οποία αυτά τα νεονικοτενοειδή να τα κρίνει επιβλαβή για τις μέλισσες. Εγώ σας λέω να δούμε τα γεγονότα τα επιστημονικά γεγονότα. Και εγώ στηρίζω την αντίρρηση της κυρίας Γκιόλιν. θα πει αυτό. Κύριο Σφαιρία. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος σε ό,τι αφορά αυτό το φάκελο και την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης. Δεν υπάρχουν ακόμα επαρκείς ε, μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν ότι εν λόγω ενεργές ε, ουσίες ε, έχουν αρνητικό αντίκτυπο αλλά ε, βλέπουμε ούτω ή άλλω δραστική μείωση τη χρήση των σχετικών ενεργών ουσιών. Ε, και δηλαδή για παράδειγμα λόγω των ε, πυρκαγιών και λόγω γενικά του κορεσμού τη χρήση των παριστοκτών στην Γεωργία. Οπότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε την επιβίωση της γεωργία μα, οπότε θα πρέπει να επιτρέπουμε αποτελεσματικά προϊόντα. Παρ' όλα αυτά, ε, υπάρχει ε, το γεγονός ότι από τη μία πλευρά δεν έχουμε ε, επαρκείς μελέτες, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να κατησχίσει η αρχή της πρόληψης και γι' αυτό θα ήθελα να απορριφθεί η, αύριο στην ψηφοφορία αυτή η έκθεση της συναδέλφου Γκέρλινγκ. Και αλλού έχει, έχει βέβαια λάβει χώρα η απαγόρευση των νοικοτινοειδών μετά, όμως από την ύπαρξη σχετικών μελετών. Οπότε εμείς στο Τη προπαρασκευαστική συζήτηση που είχε γίνει μα είπε ότι ε, όταν για παράδειγμα ε, μπαίνει το αυτοκίνητό τη ε, και κάνει μια διαδρομή μέσα από καλλιέργειε, ε, δεν υπάρχουν πια έντομα τα οποία να χτυπάνε στο μπαμπρίζ. Ε, Αντιθέτω, στη δική μου χώρα όμω, ωστόσο, εμεί βλέπουμε να υπάρχουν πολλά έντομα, χωρί να υπάρχει κανένα πρόβλημα για τι καλλιέργειε μα. Οπότε, εμεί αύριο θα καταψηφίσουμε χωρί καμία πραγματικά τύψη στη συνείδησή μα αυτή την εκθέση. Ευχαριστώ. Η κυρία Χαουτάλα. Ε, ο κύριος Χαουτάλα, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι και αυτή μια συζήτηση, λέει Σαϊτεμά, που έχει να κάνει με την επιστήμη και τους επιστήμονες. Είναι, πιστεύω, πολύ σημαντικό να ακολουθούμε μια διαδικασία. Η ΕΦΣΑ βουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πυρογνώμονες για το κατά πόσο είναι ασφαλής ή όχι χρήση. Γι' αυτό και τίνω να ακολουθώ τη δική τους τη γραμμή. Έχω όμως κάποιες ερωτήσεις επί της διαδικασίας και κάποιες ερωτήσεις που αναφέρονται και στη, στο κείμενο της κυρίας Γκέρλινγκ. Το ένα είναι η όλη αυτή συζήτηση για τον οδηγό για τις μέλισσες. Θα μπορούσε να μας πει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτροπή, ΕΦΣΑ, χώρες μέλη αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται αναθεώρηση κάποιων στοιχείων του εγγράφου αυτού. Πόσο μακριά πάει το πώς επηρεάζει την στάση μας απέναντι στα νεονικοτινοειδή. Έπειτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έκθεση λέει ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων και την μείωση του πληθυσμού των μεσηλών. Μελισσόν, το κοιτάει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοιτάει δηλαδή με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται τα φυτοφάρμακα ή κοιτάει μόνο ποια φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται και από τι αποτελούνται και δεν κοιτάει καθόλου, παραβλέπει εντελώ το θέμα του πώς αυτά χρησιμοποιούνται, με ποιο τρόπο. Και ποια είναι η λογική αυτή για το να έχουμε καλλιέργειες ε, που δεν προσελκύουν τις ε, μέλισσες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιχάουτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν συγχαρητήρια στη Τζούλη Γκέρλινγκ, η οποία δραστηριοποιείται και στις αντιρρήσεις των εφαρμοστικών πράξεων. Γιατί όταν το κάνω εγώ με επέκρινε. Τώρα βλέπω ότι αντιλαμβάνεται και εκείνη την αξία που έχει η διαδικασία αυτή. Το λέω ειλικρινά ότι χαίρομαι. Και χαίρομαι επίσης που κάνετε σαφή διάκριση ανάμεσα στο ρόλο της ΕΦΣΑ που αξιολογεί τον κινδύνο και την Επιτροπή η οποία παίρνει τις αποφάσεις γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι πρέπει να ακολουθούμε την εύσα τυφλά. Όμως η Τζουλή Γκέρλαν κάνει εδώ τη διάκριση, γιατί αυτή τη διάκριση μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες συζητήσεις που θα κάνουμε αργότερα. Έρχομαι τώρα στο περιεχόμενο. Η Τζούλη Γκέρλινγκ λέει ότι κάποιοι καθοδηγούνται από την ιδεολογία. Ωραία. Αναγνωρίζω. Υπάρχουν όμω και άλλε ιδεολογίε εκτό από αυτέ την οποία αναφέρεται, η κύριε Γκέρλινγκ. Γιατί α δούμε τα συμπεράσματα τη ΕΦΣΑ, τον Ιανουάριο, του 2013 που μιλάει για ψηλούς κινδύνου και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει το Μέο του 2013 και υπόσχεται ότι θα έρθει με αξιολόγηση βάση επόμενων δεδομένων που θα έχουμε τα επόμενα δύο χρόνια. Άρα πρέπει να κάνει κάτι. Η ΕΦΣΑ κάνει και άλλες έρευνες. Γιατί από την απαγόρευση του 2013 δεν ήταν για τις χειμερινές καλλιέργειες, ήταν μόνο για τις θερινές και δείχνει και το ολοκλήρωσε αυτό η ΕΦΣΑ και φτάσαμε στο 2016 και λέει ότι υπάρχουν κίνδυνοι και για τις χειμερινές καλλιέργειες. Οπότε βάσει αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί την αρχή της προφύλαξης. Κάποιοι εκεί που λένε ότι παρόλα αυτά υποστηρίζουν ε, την ένσταση, μαν είσαστε υπέρ της αρχής της προφύλαξης, ε, τότε δεν έχει νόημα να υποστηρίζετε την αντίρρηση, θα πρέπει να υποστηρίζετε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ λοιπόν έχω την αίσθηση ότι η αντίρρηση είναι περισσότερο ιδεολογική παρά επιστημονολογική. Πρόεδρος, κύριος Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για δύο πράγματα. Πρόκειται για την απόφαση κατά πόσον θα απαγορευτούν τα νεονικοτονοειδή και ε, άλλες ουσίες που περιλαμβάνουν ε, κατ' ουσίαν αυτά τα νεονικοτονοειδή. Αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να περιμένουμε επιστημονικές μελέτες και τα απορίσματα της ΕΦΣΑ. Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι να είμαστε αντικειμενικοί. Αντικειμενικοί όσον αφορά ε, όλες αυτές τις εξελίξεις. Ε, φοβάμαι ότι η συζήτηση είναι συναισθηματικά φορτισμένη. Κάποιοι λένε ότι θα υπάρχουν απόλυες για τη Γεωργία με συνέπειες και απόνερα. Ε, κύριος Φλόρενς έθιξε το θέμα αυτό, αλλά και άλλοι. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε αντικειμενική στάση. Δεν μπορούμε να λάβουμε απόφαση με βάση το συνέστημα. Πρέπει να λάβουμε μία απόφαση που θα στηρίζεται στην πραγματικότητα, στα επιστημονικά πορίσματα και είμαστε και υποχρεωμένοι να λάβουμε απόφαση μία λογική απόφαση. Αυτό περιμένουν από εμάς, από την Επιτροπή μας. Και ανάλογα να ψηφίσουμε και αύριο. Είμαστε υποποίηση ανάμεσα σε συμπληγάδες και τίτλε λοιπόν το εξής ερώτημα. Η φωνή των ΜΚΟ είναι εξίσου σημαντική όσο και η φωνή των παραγωγών αυτών των νησιών ή εκείνων που τις χρησιμοποιούν. Κατ' ουσίαν αυτό είναι το δίλημα που αντιμετωπίζουμε. Ακούσαμε τα υπέρ και τα κατά. Και τώρα είμαστε εμείς η Επιτροπή που πρέπει να αποφασίσει. Ευχαριστούμε κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Χαίρομαι που ακούω ότι στην Πορτογαλία υπάρχουν πολλές μέλισσες, γιατί στις χώρες μέλη από ό,τι φαίνεται δεν συμβαίνει αυτό στις περισσότερες. Και όντως έχουν μεγάλη σημασία οι μέλισσες για την γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν και τώρα και στο μέλλον. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τις απικίε των μελισσών. Γιατί έχουν να κάνουν με αυτό που τρώμε. Άκουσα πολλά για επιστημονικά πορίσματα, μελέτες και τα και υπάρχουν όντως που δείχνουν, για παράδειγμα, ότι τα νέα νοικοτινοειδή δεν καταστρέφουν μόνο τις μέλισσες, αλλά και τις πεταλούδες και πουλιά και διάφορα έντομα. Είναι από, την, από πανεπιστήμια, από Greenpeace ε, και λοιπά, σε διάφορες χώρες και έτσι αντιλαμβανόμαστε ε, γιατί μειώνονται οι απικίες των μελισσών. Γιατί ακριβώς βρίσκονται σε καλλιέργειες τις οποίες ψεκάζουμε με νέο νοικοτινοειδή. Έπειτα, έχει σημασία να λάβουμε υπόψη μας και αυτά που λέει η Εύσα. Όταν μιλάει για υψηλό κίνδυνο για τις μέλισσες, ε, σημαίνει ότι όντως μπορεί να υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Και μάλιστα ο, μπορεί να μην είναι η μόνη αιτία τα νεονικοτινοειδή για την καταστροφή των πληθυσμών της μέλισσας, αλλά σίγουρα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα. Γι' αυτό και απαγορεύει τις ε, τρεις αυτές ουσίες για να προστατευτεί ο πληθυσμός των ε, μελισσών στην Ευρώπη. Και πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί δεν μπορεί να λέμε «Α, είναι ένα αναγκαίο κακό και άρα θα αντισδεχόμαστε». Στη Γεωργία, ακόμα και αν ξέρουμε ότι πρόκειται για ψηλού κινδύνου ουσίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να τοποθετηθεί με ισχύ απέναντι σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Παίρνετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω λέγοντας πρώτα απ' όλα ότι έχει δίκιο η κυρία Κέρλιν ότι οι αντιρρήσεις πρέπει να έχουν ε, να κάνουν με την υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ισχύει όμως αυτό. Εμείς δρούμε στα πλαίσια της εντολής μας. Ο κύριος Έκχαουτ είπε επίσης ότι όταν υιοθετήθηκε ο περιορισμός των ανοικοτονιδών έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία για όσους εξακολουθούσαν να τα χρησιμοποιούν και να αποδείξουν ότι χρησιμοποιούνται με ασφάλεια. Τα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ έδειξαν όμως τώρα ότι η χρήση αυτή που εμείς απαγορεύουμε δεν είναι ασφαλής και γι' αυτό δρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναθωρεί τον παλιό περιορισμό μη εγκρίνοντας πλέον τη χρήση φυτοφαρμάκων που δεν θεωρούνται πλέον ασφαλή. Η κυρία Κέρλινγκ αναφέρθηκε επίσης και στη μελέτη του Κοινού Συμβουλίου Έρευνας. για την δράση στους επικονιαστές. Πρώτα έγινε έρευνα στους ε, γεωργούς, να δούμε πώς αντιδρούν στον περιορισμό του 2013 και τι εναλλακτική τεχνολογία χρησιμοποίησαν. Το ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικέ δεν ισχύει. Επίσης, ζητήσαμε από τους γεωργούς να σχολιάσουν για τα ωφέλη και αν έχουν επιπτώσεις από την απαγόρευση στην υγεία των μελισσών και είπαν ότι όχι καμία. Η κυρία Γκέρλιν επέκρινε ότι το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, ότι υπάρχουν κενά στη γνώση. Η αρχή της ρύθμισης είναι ότι πρέπει να αποδεικνύεται η ασφαλής χρήση και όχι το αντίθετο. Και αυτό δεν έχει γίνει. Τα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ είναι ξεκάθαρα. Πολλοί αναφέρθηκαν επίσης στον οδηγό για τις μέλισσες που χρησιμοποίησε και η ΕΦΣΑ στην αξιολόγησή της. Το πρώτο που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι το προηγούμενο σχετικό έγγραφο αναγνωρίστηκε από όλου ότι είναι ξεπερασμένο και ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αξιολογήσει σήμερα. Συνεπώς το έγγραφο της ΕΦΣΑ είναι τώρα, αυτός ο οδηγός δηλαδή, είναι η καλύτερη βάση που διαθέτουμε. Ο κύριος Χάουτεμα ρώτησε κατά πόσο αναθεώρηση του οδηγού αυτού μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις μας. Εδώ δεν είμαι σε θέση να απαντήσω, δεν μπορώ να προβλέψω μια αναθεώρηση εφόσον αυτή αποφασιστεί θα πηγαίνει. Ο κύριος Χατεμά ρώτησε επίσης και για το κατά πόσο προσελκύουν ή όχι καλλιέργειες της μέλισσες. Η ΕΦΣΑ λέει ότι η ΕΦΣΑ δεν μπορούσε να καταλήξει με βεβαιότητα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και στις περιπτώσεις τώρα που συζητάμε η ΕΦΣΑ είπε ότι υπάρχει κίνδυνος και για τις ε, επόμενες καλλιέργειες, μετά τα ζαχαρότευτλα δηλαδή. Ότι η ουσία παραμένει υδραστική στο έδαφος και μπορεί να επηρεάσει και τις επόμενες καλλιέργειες. Γι' αυτό αναφέρεται στα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ. Επίσης, κύριε Γκέρλινγκ είπε ότι θα έπρεπε να είχαμε κοιτάξει τις επιπτώσεις της καλλιέργειας, απώλεια καλλιεργειών, και να γίνουν και άλλες μελέτες αντικτύπου. Δεν προβλέπεται όμως τίποτα τέτοιο στον κανονισμό που ακολουθούμε. Αν είχαμε χρησιμοποιήσει τέτοια επιχειρήματα για την απόφασή μας, τότε θα είχαμε ξεπεράσει την εντολή μας και τις ε, εφαρμοστικές μας, εκτελεστικές μας αρμοδιότητες. Τέλος, συμμερίζομαι την επιθυμία της κυρίας Γκέρλινγκ για παρετέρω έρευνες και συμφωνούμε να γίνουν τέτοιες έρευνες για την υγεία των μελισσών. Είναι εφικτό βάσει του ορίζοντα 2020 και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα ώστε να ερευνήσουμε την υγεία των μελισσών και πώς συνδυάζεται αυτή με τη ρήπανση του περιβάλλοντος και τη χρήση φυτοφαρμάκων. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύει και σε ένα πρόγραμμα δράσης για τους επικονιαστές είπε στο τέλος, ρώτησε μάλλον, αν εμείς ασχολούμαστε μόνο με τις δραστικές ουσίες ή και με τη χρήση τους. Ναι, και με τη χρήση τους. Υπάρχει μια οδηγία για τα φυτοφάρμακα που το προβλέπει αυτό. Ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πορό να υποβάλει μια έκθεση για το αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Οπότε ναι, ασχολούμαστε και με τη χρήση και όχι μόνο με τις ουσίες αυτές καθ' Εδώ θα ολοκληρώσω, ξέρω ότι δεν έχω χρόνο, ενώ θα μπορούσα να σας πω και πολύ περισσότερα βέβαια. Πρόεδρος. Ωραία, ναι. Η κυρία Γκέρλινγκ τώρα. Σύντομα παρακαλώ. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Πρέπει να σας πω ότι δεν βγήκαν και πολλά. Άκουσα αυτά που περίμενα να ακούσω ο τόνος ήταν έτσι λίγο έντονος. Εντάξει. Θα μπορούσα κι εγώ να μιλήσω για 20 λεπτά και να απαντήσω σε όλα τα θέματα ένα προς ένα. Κάποιος μίλησε για την προφύλαξη και την υποκατάσταση. Μα δεν υπάρχει τίποτα για την υποκατάσταση εδώ. Και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την αντικατάσταση, την αναθόρηση μάλλον της οδηγίας για την προστασία των φυτών και να δούμε ποιος είναι ο αντικτυπός της. Γιατί δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι τα ζωτούχα παραμένουν στο έδαφος ή για το τι περιοχή καλύπτουν. Δεν υπάρχει τέτοια απόδειξη. Οπότε γιατί να μην καθίσουμε να σκεφτούμε και τέτοια ζητήματα. Τεχνικά μπορεί να έχετε δίκιο, δεν προβλέπετε στην νομοθεσία, θα έπρεπε όμως και θα ήθελα τα μέλη της Επιτροπής αυτής να το ζητήσουν με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως προσπαθούν να προστατεύσουν ε, τις μέλισσες ε, απαγορεύοντας τα φυτοφάρμακα. Ωραία, δεν θα τα πω όλα. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε και προσβλέπω στην ψηφοφορία. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Αύριο θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, 4 και 2 τώρα για την κοινή συνάντηση που έχουμε την Ήτρε. Ευχαριστώ.